Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Έγκριση μερίσιας διάταξης πρώτα. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Συνεπώς εγκρίνεται. Έχω κάποιες ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτη, έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2020. Για πρώτη φορά λοιπόν υπό αυτή την ε, κοινοβουλευτική θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της, ε, του ελέγχου της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Κρατική Πρεδρία οργανώνουν την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2020 που θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2020 στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα συγκεντρώνει βουλευτέ, από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υποψήφιες χώρες και παρατηρητές για να εξετάσουν οικονομικά, δημοσιονομικά και κοινωνικά θέματα. Αποτελείται από μία ολομέλεια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και από κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Προ το παρόν έχουν ε, καταγραφεί για να συμμετάσχουν 97 μέλη από 32 σώματα. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να συμμετέχετε κυρίως στι συναντήσει τη ΕΝΚΟΝ για τη φορολόγηση και τα βιώσιμα δημοσιονομικά. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευκαιρία που έχετε το Κοινοβούλιο να ενισχύσει τη δημοκρατική λογοδοσία όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Κάτι άλλο τώρα για τους κεντρικούς ε, αντισυμβαλόμενους και την ανάκαμψη και εξηγένσή του. Ο πρώτο τριμερή διάλογο έλαβε χώρα στι 28 Ιανουαρίου. Οι συνομοθέτες τόνισαν την σημαντική πρόταση αυτή στα πλαίσια τη συγκέντρωση κινδύνων με του κεντρικού αντισυμβαλόμενου μετά την δημοσιονομική κρίση. Αναγνωρίζουν ότι η θέση του διαφέρει βέβαια για πολλά σημαντικά θέματα, κυρίω όσον αφορά για το ποιο αποφασίζει το νέο πλαίσιο και ποιο τελικά είναι αυτό που πληρώνει, με ποια σειρά για να επιβιώσει ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος. Θεωρούν ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε περισσότερο διάφορα ζητήματα σε πολιτικό επίπεδο. Συμφώνησαν επίση να ξεκινήσει ο νέο τριμερή διάλογο συζητώντα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, ανάκαμψη. Για παράδειγμα, όσον αφορά το λεγόμενο skin in the game, δηλαδή πώς ε, διατηρείται το τμήμα του κινδύνου όσον αφορά του τίτλου και όσον αφορά τα περιθώρια που υπάρχουν. Αυτά, είναι, αυτά έχουν να κάνουν με τις δραστηριότητές μας και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τον νομισματικό διάλογο με την Κριστίν Λαγκάρδα, που είναι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, από τον προηγούμενο νομισματικό διάλογο που είχαμε αρχές Δεκεμβρίου, οι οικονομικές προοπτικές δεν έχουν αλλάξει πολύ. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ευθυγραμμίζονται με την συνεχιζόμενη αλλά μέτρια ανάπτυξη της ε, Ευρωζώνης. Κάτι το οποίο οφείλεται στις αδυναμίες του διεθνούς εμπορίου και σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που έχει επηρεάσει κυρίως την Ευρωζώνη, την ε, μεταποίηση κλπ. Όμως συνεχίζεται η ανάπτυξη στην, στην απασχόληση, αν ε, και αδύναμη, όπως επίσης και στους μισθούς, που βοηθούν την αντοχή της οικονομίας μας. Παρόλο ε, λοιπόν όπου υπάρχουν αδυναμίες, παρόλο αυτά υπάρχει κάποια αύξηση στον υποκείμενο πληθωρισμό που δείχνει την ε, αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Οι προσδοκίες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αλλά έχουμε είτε σταθεροποίηση είτε ενισχύσει την κατάσταση. Μεσοπρόθεσμα ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί εξαιτία των ε, πολιτικών μας, της οικονομικής ε, επέκτασης και της ανάπτυξης. Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα βασικά επιτόκια παραμένουν μετάβλητα όσο οι προοπτικές ε, του πληθωρισμού προχωρούν για να πετύχουν την σύγκληση προς και κάτω από το 2%. Θα συνεχίσει επίση την έρευνα καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματο για την αγορά στοιχείων ενεργητικού με ύψο 20 δισεκατομμυρίων ευρώ μηνιαίω. Και αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτική ε, και ότι πριν λήξουν θα συνεχίσει η αύξηση των βασικών επιτοκίων. Επίσης, θα συνεχίσει η επανεπένδυση. Ε, μας ενδιαφέρουν θέματα περιβάλλοντος, παγκοσμιοποίησης, και δομών και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει μια αναθεώρηση ή επανεξέταση τη στρατηγική τη νομισματική πολιτική που είναι από το 1998 και να διευκρινίσει ε, και διευκρινίστηκαν επίση διάφορα στοιχεία το 2003 και θα βασιστεί σε ποσοτική διατύπωση τη σταθερότητα των τιμών, την δέσμη εργαλείων νομισματική πολιτική, οικονομική και νομισματική ανάλυση και επικοινωνιακέ πρακτικέ. Υπάρχουν και άλλε παράμετρο όπω είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η απασχόληση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα που θα αποτελέσουν επίσης μέρος της επανεξέτασης. Η επανεξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί βάσει της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα, όπως αυτή αναφέρεται στη συνθήκη, και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020. Όλοι εκτιμούμε όλους ιδιαίτερος ότι έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ήδη και την προηγούμενη, στην ακρόασή σας μας αναφερθήκατε σε αυτό, όπως και στον τελευταίο νομισματικό διάλογο. Σίγουρα θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις για το πεδίο εφαρμογή και για τις επιθυμίες όσον αφορά αυτή την επανεξέταση, αλλά πιστεύω ότι εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τονίσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την επανεξέταση και κυρίως αυτή τη κοινοβουλευτική επιτροπή. Συνεπώς, σήμερα η Πρόεδρος Λαγκάρτα μα μας τις προοπτικές τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την οικονομική και δημοσιονομική ανάπτυξη και έχουμε ε, διαλέξει δύο θέματα στην Επιτροπή μας για να προετοιμάσουμε αυτόν τον διάλογο και το ένα είναι η εξολόγηση κινδύνων που έχουν να κάνουν με την ε, σταθερότητα και το άλλο είναι η επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε αποφασίσει για αυτά τα θέματα, έχουμε συζητήσει με εμπειρογνώμονε και υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλά ενδιαφέροντα λοιπόν θέματα έχουμε να συζητήσουμε και πολλέ είναι οι προσδοκίε μα από αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Συνεπώ, κύριε Λαγκάρτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι ευρωβουλευτέ τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, κυρίε και κύριοι. Καλή σα μέρα. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και πάλι ενώπιον σα μετά την πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαμε το 2020 πρόσφατα δηλαδή και κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα γενικότερα αποφάσισαν να ξεκινήσει την επανεξέταση της στρατηγικής της για την νομισματική πολιτική, για να είμαι συγκεκριμένη. 16 χρόνια πριν είχαμε μία επανεξέταση της στρατηγικής μας για την νομισματική πολιτική και των Δεκέμβριο το συζητήσαμε. Το 2003 ο κόσμος ήταν εντελώ διαφορετικός. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, το οποίο σημαίνει ότι η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουν υπάρξει δομικές αλλαγές, έχει αλλάξει το περιβάλλον και το οικονομικό, αλλά και άλλο, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ε, σε αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, οι τάσεις για μείωση της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και το δημογραφικό, όπως επίσης και η κληρονομιά που έχουμε από την οικονομική κρίση, έχουν σαν αποτέλεσμα τα επιτόκια να παραμένουν χαμηλά. Τα χαμηλά επιτόκια και ο χαμηλός πληθωρισμός έχουν μειώσει και το περιθώριο που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και άλλες κεντρικές ε, τράπεζες να χρησιμοποιήσουν συμβατικά μέτρα για την νομισματική πολιτική. Επίσης, νέες προκλήσεις, περιβαλλοντικές, ε, ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση, έχουν επίσης επηρεάσει την εξέλιξη των τιμών και έτσι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ελέγχουν την κατάσταση οι, Ευρωπαϊκές, οι Κεντρικές Τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επηρεάζουν βέβαια την πολιτική. Υπό το φως των αλλαγών αυτών τώρα ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε σε αυτήν την επανεξέταση ώστε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να φέρουμε σε πέρα στην εντολή μας προς το καλύτερο συμφέρον των Ευρωπαίων. Την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, σας υποσχέθηκα ότι θα ακούσω τον κόσμο. Θα προσπαθήσω να καταλάβω καλύτερα τις ανησυχίες τους και μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, διάβασα διάφορα έγγραφα που ετοιμάσατε όσον αφορά την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την ευαισθησία που δείχνει ο κόσμος για τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εννοείται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας θα είναι κατά πρώτο λόγο αυτός που θα συμμετέχει στο διάλογο αυτό και θα εφαρμόσουμε την αρχή της αμφίδρομης επικοινωνίας όπως υπογράμμισα και στην προηγούμενη συνάντησή μας. Συνεπώς χαίρομαι πάρα πολύ που μου ζητήσατε να έρθω εδώ να συζητήσω μαζί σας το θέμα της επικοινωνίας της ΕΚΤ σήμερα. Πρώτο όμως επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ποια είναι η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη και δεν θα διαφέρει πολύ από αυτά τα οποία είπατε κι εσείς ε, μόλις κυρία Πρόεδρε. Συνεπώς, βάσει των προσδοκιών μας, η οικονομία της Ευρωζώνης συνεχίζει να αναπτύσσεται αλλά με χαμηλό ρυθμό. Η εσωτερική οικονομία ε, παραμένει ανθεκτική. Η ιδιωτική κατανάλωση, για παράδειγμα, αύξησε, αυξήθηκε 0,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2019 και υπάρχουν και άλλες βελτιώσεις στις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Η ανεργία βρίσκεται στο 7,4%, κάτι που είναι το χαμηλότερο ε, ποτέ από τον Ιούλιο του 2008. Οι άνεργοι αυξάνονται και είναι 11 εκατομμύρια. Εσωτερικά διαπιστώνουμε ότι σε πάρα πολλούς τομείς υπάρχει ε, βελτίωση. Παρ' όλα αυτά, παράγονται σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης. Οι διάφοροι δείκτες δείχνουν ότι η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, όπως δείχνει και ο δείκτης για τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, που βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση πέντε συνεχόμενους μήνες από τον ε, Ιανουάριο και τους προηγούμενους 18 μήνες. Υπάρχουν βεβαιότητες βέβαια όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, για παράδειγμα, αλλά ευτυχώ οι εντάσεις αυτές μειώνονται. Υπάρχουν όμως άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι παραμένουν, όπως επίσης το θέμα του κορονοϊού και άλλες ανησυχίες. Οι γενικές επιδόσεις καθυστερούν την μετακύληση της αύξησης των μισθών, για παράδειγμα, στις τιμές και στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός που υπολογίζεται από τον αναρμονισμένο δίκτυο τιμών καταναλωτής ήταν 1,4% το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις προσδοκίες μας και σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τους προηγούμενους μήνες. Η οικονομία της Ευρωζώνης συνεχώς συνεχίζει να απαιτεί στήριξη από την νομισματική μας πολιτική, η οποία αποτελεί μια ασπίδα προστασίας. Βλέπουμε ότι οι πολιτικές μας εξαρτώνται και από τις οικονομικές κατάστασεις στην πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επίπεδα δανεισμού για τις επιχειρήσεις είναι 10 μονάδες βάσης κάτω από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Και για τα νοικοκυριά, για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, βρισκόμαστε σε 40 μονάδες κάτω και σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι θετικές συνθήκες χρηματοδότησης ενισχύουν τις επενδύσεις και τις δαπάνες των καταναλωτών στην Ευρωζώνη παρά τις αρνητικές εξελίξεις στην παγκόσμια ζήτηση. Συγχρόνως όμως συνεχίζουμε να ελέγχουμε στενά τις ε, παρενέργειες των μέτρων αυτών. Τα χαμηλά επιτόκια έχουν πολλά ωφέλη για την οικονομία στην Ευρωζώνη. Όμως, το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης ενθαρρύνει περισσότερο δανεισμό και περισσότερους κινδύνους από μη τράπεζες όπως είναι χρηματοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία και συνταξιοδοτικά ταμεία. Επιπλέον οι αγορές ακινήτων σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης αυξάνουν τις τιμές παρά τα χαμηλά επιτόκια, γιατί αυτά είναι ένας μόνος παράγοντας που συμβάλλει στην απόφαση κάποιου να επενδύσει σε κίνητα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι αρχές χρησιμοποιούν μακροπροληπτικά μέτρα στοχευμένα για να μειώσουν τους κινδύνους και να πετύχουν τη σταθερότητα. Συγχρόνως δημοσιονομικές και δομικές ε, πολιτικές έχουν να παίξουν ρόλο μέσα σε ένα κλίμα χαμηλών επιτοκίων βοηθούν και ενισχύουν την ε, παραγωγικότητα. Έτσι, στηρίζονται επίσης και τα δικά μας νομισματικά μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τώρα επιτρέψτε μου να έρθω στο θέμα της επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για όσου από εσά παρατηρείτε τι γίνεται στι κεντρικέ τράπεζε, θα έχετε διαπιστώσει ότι έχουν διανύσει πολύ δρόμο όσον αφορά την επικοινωνία του. Τα διάφορα όργανα, όπω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν προσπαθήσει να δίνουν περισσότερε πληροφορίε και να εξηγούν καλύτερα την πολιτική μα για να ανταποκρίνονται και στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του κοινού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικό σας κοινοβούλιο δηλαδή, έχει ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ακολουθήσει αυτό το δρόμο από την αρχή. Ένα από τα θέματα τα οποία έχουν επιλεγεί για την πρώτη συνάντηση ΕΚΟΝ το 1999 ήταν η πολιτική επικοινωνίας και διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε η καλή επικοινωνία αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την νομιμότητά μας απέναντι στον κόσμο, τον οποίο εξυπηρετούμε. Οι κεντρικοί τραπεζίτες το ξέρουν ότι είναι προς όφελός μας η καλή επικοινωνία. Να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε ξεκάθαροι είναι πολύ βασικό προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές στις δικές μας οι πολιτικές. Να σταθμίζουμε καλά την επικοινωνία μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα τις ενδείξεις που σας ε, δίνουμε και στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς. Αποτελεί ένα εργαλείο της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας. Παραδοσιακά, ως κεντρικοί τραπεζίτες, νιώθουμε πιο άνετα όταν συζητάμε με εμπειρογνώμονες και με αγορές από ό,τι όταν μιλάμε με το ευρύ Οι αγορές παρακολουθούν τη δράση μας, παρακολουθούν τα όσα λέμε, τα όσα δεν λέμε και μελέτες ε, δείχνουν ότι γενικά μας καταλαβαίνουν καλά. Είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί επίσης για το πώς οι αγορές ερμηνεύουν ή παρερμηνεύουν τη δράση μας. Όμως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην επικεντρώμαστε μόνο στην επικοινωνία αυτή με τις αγορές και δημιουργούμε το δικό μας ε, σύστημα, κλειστό σύστημα. Και αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και η εκρόση που είχα εδώ ενώπιόν σας είχα πει ότι η Προεδρία μου θα φροντίσει να καλύψουμε και να δημιουργήσουμε γέφυρες με το κοινό. Οι δικέ μα έρευνε δείχνουν ότι πολλοί Ευρωπαίοι έχουν ακούσει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά πολύ λίγοι αντιλαμβάνονται πραγματικά τι κάνουμε. Και σίγουρα όχι γιατί το κάνουμε ή πώς εξυπηρετεί το κοινό καλό το έργο μας. Και αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Όχι απλώ για να είμαστε δημοφιλείς, δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά ώστε οι Ευρωπαίοι να καταλαβαίνουν τι κάνουμε και πώς το κάνουμε προς όφελός τους. Επίσης, ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε μια νέα έρευνα ε, βάσει της οποίας ζητάμε τους καταναλωτές ποιες είναι οι δικές τους προσδοκίες όσον αφορά τον πληθωρισμό, όσον αφορά τη στέγαση, όσον αφορά την κατανάλωση, όσον αφορά την αποτεμίευση και την αγορά εργασίας. Πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα τη σχέση αυτή και οι καταναλωτές πρέπει να μας καταλαβαίνουν καλύτερα, ομάδες της κοινωνίας, ε, υπάρχουν διαφορές οι άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο ή στην πόλη. Οι καθημερινές αποφάσεις όμως των επιχειρήσεων και των ανθρώπων επηρεάζονται από τη δικιά μας την πολιτική και, τις δικές μας, ε, και τη δικιά μας επικοινωνία. Συχνά η γλώσσα μας είναι σκοτεινή, δεν την αντιλαμβάνεται ο κόσμος και η πολιτική μας θα είναι λιγότερο αποτελεσματική, όπως επίσης και τα αποτελέσματα του έργου μας κινδυνεύουν αν ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί περισσότερο και θα αντιληφθεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν τη δικιά τους τράπεζα αν καταλαβαίνει τις αποφάσεις μας, γιατί έχουν σημασία για αυτούς και πώς επηρεάζεται η καθημερινότητά τους από αυτές. Και γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η επανεξέταση της στρατηγικής μας που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο στην τελευταία μας συνεδρίαση θα εξετάσει και την επικοινωνία μας. Η επικοινωνία εκλαμβάνεται πολλές φορές σαν μονόδρομος, με πολλές προσπάθειες σε μηνύματα τα οποία παρουσιάζουμε. Όλοι επικεντρωνόμαστε στο να μιλάμε, στην ομιλία μας. Μας αρέσει να μιλάμε, να ακούμε τη φωνή μας. Όμως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να επικεντρωθούμε εξίσου και στο να ακούμε, να ακούμε τον κόσμο. Και όπως ο Τζον Μάρσαλ έχει ήδη πει, ήδη από το 1800, το να ακούει κανείς ε, καλά είναι εξίσου σημαντικό ως επικοινωνία, όπως και το να μιλάει καλά. Έτσι έχουμε δύο αυτιά, ένα στόμα, θα πρέπει όλα να τα χρησιμοποιούμε εξίσου. Γι' αυτό λοιπόν ένα στοιχείο βασικό της στρατηγικής μας θα είναι να συμπεριλάβουμε το στοιχείο ακριβώς αυτό. Να ακούμε δηλαδή και αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας και διαρθρωτικά. Ήδη ο διάλογος με τη δικιά σας επιτροπή είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά επιπλέον εγώ έχω υπόψη μου και διάφορες άλλες ε, ενέργειες και δράσεις που θα λάβουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αποκινούμε τους συναδέρφους μας από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, ώστε ολόκληρο το ευρωσύστημα να συμπεριληφθεί και ο διάλογος αυτός να γίνεται και στη γλώσσα του καθενός, στις εθνικές γλώσσες δηλαδή, στις διάφορες χώρες. Θέλουμε να ακούσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, τους ακαδημαϊκούς, το χρηματοπιστωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της, φοιτητέ και πάρα πολλοί κόσμο από διάφορες κατηγορίες. Η πρώτη τέτοια δράση θα λάβει χώρα εδώ τέλη Μαρτίου στις Βρυξέλλες και ελπίζω να έχω εκπροσώπους και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εδώ, από τα ευρωπαϊκά όργανα και θα προσκληθείτε κι εσείς όλοι να συμμετάσχετε εφόσον το επιθυμείτε. Επίσης θα έχουμε και ένα πόρταλ online όπου όλες οι πληροφορίες όσον αφορά την επανεξέταση της στρατηγικής μας θα είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό και όσο γίνεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ήδη γίνεται πολλή δουλειά και θα δούμε ότι θα έχουμε και τη δημοσίευση πολλών ε, γράφων και πληροφοριών. Μέσω αυτών των διάβλων θέλουμε να μάθουμε από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από τον κόσμο που τις εκπροσωπεί. Τι τους νοιάζει περισσότερο. Οι τιμές, τη στέγαση, η αβεβαιότητα, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση. Ποια είναι η γνώμη τους. Και θέλουμε να αξιολογήσουμε πώς τις ανησυχίες αυτές μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη μας στις δικές μας δράσεις και την επικοινωνία μας, πάντα στα πλαίσια της εντολής μας. Συνεπώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, η επανεξέταση που μόλι ξεκινήσαμε θα είναι σε βάθο. 11 μήνε θα μα απασχολήσει ο διάλογο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα είναι σε βάθο. Οι τακτικέ ακροασει εδώ στην ΕΚΟΝ θα αποτελέσουν και τη σπονδυλική στήλη των συζητήσεων αυτών που δεν θα περιοριστούν όμω μόνο σε αυτές τις ακροάσεις. Θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε να συνεχίσουμε το διάλογό μα σύντομα. Προσβλέπω σε συνάντηση, επίσκεψη της αντιπροσωπείας της δικιάς σας επιτροπής τώρα τη Δευτέρα στη Φραγκφούρτη και θα σας ξανασυναντήσω την Τρίτη στο Στρασβούργο. Την επομένη. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η επικοινωνία μας εντείνεται αυτές τις μέρες με όλου εσά και του συναδέρφους σας. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τώρα περιμένω τι ερωτήσει σα, όπω το επιθυμείτε κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε τώρα με τις ερωτήσεις ε, με τον γνωστό τρόπο. Πέντε λεπτά για ερώτηση και απάντηση. Ξεκινάμε με τον Μάρκους Φέρμπερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ε, κυρία Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω στα γερμανικά. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην εξέταση της νομισματικής ε, πολιτικής μέλος ε, του αρμόδιου διευθυντηρίου αναφέρθηκε στους διάφορους ε, παράγοντες ε, που επηρεάζουν την ασθενή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οπότε τίθεται το ερώτημα εάν είστε σε θέση να πετύχετε τον στόχο που έχετε θέσει οι ίδιοι, δηλαδή κοντά αλλά όχι ακριβώς 2% όταν και η ανάπτυξη θα είναι κάτω από το 2%. Θα δούμε λοιπόν πώς ε, θα μπορέσουν να συμβαστούν οι προσδοκίες για την ανάπτυξη με τις προσδοκίες για τον ε, πληθωρισμό και υπάρχει η τελευταία Financial Stability Review από τον Νοέμβριο που μιλήσατε για αύξηση των ε, κινδύνων δηλαδή οι κίνδυνοι αυξάνονται αν διαβάζω καλά και θεωρώ πως αρκετοί από αυτού του κινδύνου ε, συνδέονται με τα χαμηλά επιτόκια. Δηλαδή η χαλαρή νομισματική πολιτική αυξάνει την τιμή των διαφόρων ε, στοιχείων ε, ενεργητικού. Απ' την άλλη πιέζει την κερδοφορία των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν το ερώτημα είναι πώς βλέπετε την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μπορεί να αντιδρά σε αυτό το περιβάλλον εάν υλοποιηθούν τελικά αυτοί οι κίνδυνοι. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Δύο πράγματα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω. Πρώτον, η αναθεώρηση της στρατηγικής μας θα εξετάσει όλες τις πτυχές της νομισματικής πολιτικής ε, και θα πάρει χρόνο. Δηλαδή έχουμε θέση ως ε, προθεσμία το Δεκέμβριο του 2020 για την ολοκλήρωση. Πριν από αυτό όμως θα έχουμε συνεδριάσεις του ΔΣ που θα εξετάσουν την νομισματική πολιτική και θα αποφασίσουν ε, με βάση τους αριθμούς τα στοιχεία την νομισματική μας πολιτική. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτό να το κάνουμε με βάση τις υφιστάμενες αρχές ε, και κριτήρια μέχρι να ολοκληρωθεί όπως είπαμε η επανεξέταση αυτή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ακάθεκτη την, ε, τον κανονικό καθορισμό της ε, νομισματικής μας πολιτικής. Λοιπόν, βεβαίως πρέπει να δούμε όλα τα αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τον αντίκτυπο που είχε και έχει και αν δούμε τον αντίκτυπο που έχει το γεγονός ότι έχουμε περιλάβει ε, στο συμβατικό και μη συμβατικό επίπεδο διάφορα εργαλεία ε, νομίζω ότι είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα αναφερόμαστε συνεχώς στη δημιουργία θέσεων εργασίας δεν θα αναφερθώ τώρα στα 11 εκατομμύρια ε, θέσει εργασία ε, που δημιουργήθηκαν από το 2013 γιατί η νομισματική πολιτική ήταν ένας παράγων. Αλλά σαφώς η νομισματική πολιτική ε, μπορεί να πει ότι έχει ένα μερίδιο στην δημιουργία αυτών των θέσεων εργασία. Μπορεί επίσης να πει ότι έχει συνεισφέρει στην αυξημένη ανάπτυξη από το 2013 και στο ίδιο πνεύμα έχει συνεισφέρει και στην αύξηση ελαφρώς του πληθωρισμού. Ε, κατά τη διάρκεια των ετών αυτών. Οπότε πρέπει να δούμε τι και αποτελέσματα και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις, τη ζωή των ανθρώπων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να πούμε ότι έχει υπάρξει αποτελεσματική. Υπάρχουν βεβαίω και αυτά τα οποία αναφέρατε αν έχει αυτές τις παρενέργειες και να το δούμε από τη σκοπιά κόστους-οφέλους ε, των θετικών και των δυνητικά άλλων ε, αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής. Εγώ δεν θα έβγαζα το συμπέρασμα ότι η νομισματική μας πολιτική ήταν ο βασικός παράγων στην αύξηση των τιμών των ακινήτων ή της πτώσης της κερδοφορίας κάποιων τραπεζών στην Ευρωζώνη. Ίσως να έχει συνεισφέρει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δεδομένο γιατί αν το συγκρίνουμε με άλλα περιβάλλοντα όπου ήταν χαμηλά τα επιτόκια ε, δεν είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Επίσης, δεν θα έλεγα ότι οι τιμές των σπιτιών και των ακινήτων έχουν αυξηθεί γενικά. Είναι τελείως διαφορετική η εικόνα στην Ευρωζώνη, αν δούμε τις πόλεις και την Ήπεθρο και όπως είπα και στην αρχική μου δήλωση δεν ε, οφείλεται εντελώς ε, στα επιτόκια και στο πολύ χαμηλό κόστος ε, χρηματοδότησης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά παρακολουθούμε και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις παρενέργειες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Χώνες Φερνάντες από τους Σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Θα μιλήσω ισπανικά. Πριν από λίγου μήνε, όταν ήρθατε σε αυτή την επιτροπή στη διαδικασία διορισμού για να εκλεγεί ο νέο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σα ρώτησα με εκείνη την ευκαιρία για τη δυνατότητα να ξεκινήσει αυτή η επανεξέτηση του στρατηγικού πλαισίου ε, δράσεις για την ε, νομισματική πολιτική και βλέπω ότι ο θεσμός σας ε, το ξεκίνησε και θέλω να σας συγχαρώ που ξεκινήσαμε θέλω, αυτή τη συζήτηση. Αυτή λοιπόν η συζήτηση που μόλις ξεκίνησε για την επανεξέταση της νομισματικής πολιτικής νομίζω πως υπάρχει ένα κομμάτι για την επικοινωνία που εσείς πολύ ωραία το εξηγήσατε στη σημερινή σας εισήγηση αλλά θα ήθελα να σας ε, επιστήσω την προσοχή σε αυτή την πορεία γιατί είναι βέβαιο και το είπατε και εσείς ότι πρέπει και οφείλουμε να εξηγήσουμε καλύτερα τις πολιτικές ε, της ε, ΕΚΤ να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες όμως είναι αλήθεια πως η ΕΚΤ από τη φύση της επειδή πρέπει να είναι ανεξάρτητη δεν μπορεί να είναι αντικείμενο καθημερινή συζήτηση στα σπίτια και στις συζητήσεις στις κουβέντες των πολιτών, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί έτσι να χάσουμε τον ανεξάρτητο χαρακτήρα, την αυτονομία του θεσμού αυτού. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Σας συγχαίρω που ναι θέλετε και χαίρομαι για αυτή σας την ε, πρόθεση να επικοινωνήσετε καλύτερα, αλλά είναι και θέμα ε, εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται όταν ε, κανείς είναι πιο κοντά στο κοινό, αλλά είναι λίγο εκτός της καθημερινής πολιτικής συζήτησης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά ήθελα να σας πω, αυτή την ανησυχία μου να μοιραστώ μαζί σας. Τώρα, όσον αφορά την επανεξέταση των στόχων και των μέσων της νομισματικής πολιτικής, τις τελευταίες μέρες διεφάνει δυνατότητα να ενταχθεί στον δίκτυο πληθωρισμού Η πιθανότητα, ιδιαίτερα για κάποια ενεργά στοιχεία του τα θέματα στέγασης να μπει μέσα στις τιμές του πληθωρισμού. Πιστεύω πως πρέπει αυτό να το επανεξετάσουμε ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη συμμετρία. Αν υπάρχουν προβλήματα γιατί μπορούμε να μην φτάσουμε στο 2% όπως έλεγε ο συνάδελφος Φέρμπερ και άρα τότε πρέπει να δουλέψουμε πάνω στον δίκτυο για να βάλουμε τα δύο αυτά, ε, τις δύο αυτές μονάδες, ε, ε, εντάξει. Έπειτα, Επίσης, για να αποφύγουμε τις παράπλευρες ε, επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, ε, επιρροή δηλαδή στη φορολογική πολιτική και θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας για τη χτεσινή ανακοίνηση της ε, Κομισιόν πάνω σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα, κυρία Λαγκάρντα. Σας ευχαριστώ πολύ και όσον αφορά τη σύστασή σας για την επικοινωνία, την οποία θα λάβω σοβαρά υπόψη και για την ερώτησή σας όσον αφορά τα κόστη ε, στέγασης. Για την επικοινωνία καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε και νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να προχωράμε με προσοχή, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να ακούμε όσο γίνεται περισσότερο καθώς θα δίνουμε βάση και θα ακούμε περισσότερο, θα χρειάζεται κάπως να εξηγήσουμε και το τι ακριβώς κάνουμε, γιατί για μένα ήταν έκπληξη που όταν είδα πόσα λίγα ξέρει ο κόσμος για την ε, ΕΚΤ και τι ακριβώς κάνει. Και όταν μιλάμε για το ευρωσύστημα βλέπετε να γουρλώνουν τα μάτια και να απορούν. Τι τούτο σκέφτεται ο κόσμος. Όμως νομίζω το οφείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ε, να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε και γιατί έχει σημασία το τι κάνουμε εμείς. Γιατί εμείς είμαστε οι ε, θεματοφύλακες του νομίσματος πώς και γιατί είμαστε εμείς ένας ενοποιητικός παράγοντας στο ευρώ, πάει καλά και είναι σεβαστός σε όλη την ευρωζώνη. Πιστεύω πως και γιατι ειμαστε εμεις ενας ενοποιητικο παραγοντας στο ευρω παει καλα και ειναι σεβαστος ολη την ευρωζωνη πιστευω πως αυτο πρεπει να το κάνουμε και θέλουμε, όπως σας είπα, να ακούσουμε τους πολίτες. Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να προχωράμε με προσοχή και να μην αυξήσουμε υπερβολικά τις προσδοκίες, καθώς και να μην αφήσουμε κανέναν ε, να νομίσει ότι μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα από όσα <laughs> στην πράξη είναι δυνατόν. Δεν Πιστεύω το θέμα της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας είναι ακριβώς κάνε αυτό που λες, αλλά μην το ξεπερνάς, μην λες παραπάνω, γιατί όταν είναι υπερβολικά ψηλές οι προσδοκίες ακολουθεί απογοήτευση και κατά συνέπεια και δυσπιστία. Για το θέμα της ε, στέγασης. Για την ώρα το HACP μετρήσεις ε, ε, δηλαδή πληθωρισμού στην Ευρώπη δεν λαμβάνει υπόψη το οικιστικό κόστος ε, όταν κανείς είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου. Από ό,τι θυμούμε, σε ολόκληρο το δίκτυ το οικιστικό κόστος αντικατοπτρίζει το 6,5 του συνόλου του κόστους. Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε, οικογένεια, φίλους κτλ, 6,5% είναι μάλλον λίγο για ε, να μην πω πολύ λίγο. Πώς ανταποκρινόμαστε λοιπόν σε αυτό χωρίς να κατηγορηθούμε και χωρίς να διατρέξουμε τον κίνδυνο ότι αλλάζουμε τους στόχους. Γιατί ε, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή μετράς για κάποια περίοδο σε σύγκριση με συγκεκριμένη δομή και τώρα αποτείνεις αλλαγή αυτής της δομής. Το ίδιο νομίζω πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, το τι θεωρεί ο, ο κόσμος ως δομή κόστους. Εάν το οικιστικό κόστος είναι τόσο χαμηλό, θα πρέπει αυτό να το αφισβητήσουμε και να δούμε κατά πόσο αυτό είναι θεμητό ή όχι. Επιπλέον, θα πρέπει, ε, θα αντιμετωπίσουμε μάλλον δυσκολίες όσον αφορά την αξία της ε, ε, χρήσης ενός ε, ακινήτου του οποίο είσαι ιδιοκτήτης και το πώς η αξία του ε, μεταβάλλεται, αυξάνεται, μειώνεται σε σχέση με την αρχική επένδυση. Αυτό νομίζω οφείλουμε να το κάνουμε ώστε να σκεφτούμε το πραγματικό κόστος και πώς αυτό αντικατοπτρίζεται. Να θέσουμε δηλαδή τα βασικά ερωτήματα για το πώς μπορούμε καλύτερα να το αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τις αρχές αλλά και τις πραγματικές δαπάνες του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν περάσουμε στον επόμενο μιλητή, παρακαλώ, σας υπενθυμίζω, πέντε λεπτά είναι η κάθε έρωτα οπότε δύο λεπτά για την ερώτηση μόνο για να μπορεί και η κυρία Λαγκάρντ να σας απαντάει εκτενώς, αλλά να μπορέσουν και όλο να πάρουν το λόγο. Κύριος Λουίτ Γκαργκάνο. Κυρία Λαγκάρ, ναι, 1993 είπατε ήταν η πρώτη φορά που είδα στην Eurostat τον δείχτη αυτό ότι μόν καταναλωτή. Ε, χρόνια πίσω βέβαια. Τι μου θυμήσατε. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει αρκετά για να αντιμετωπιστεί η τραπεζική κρίση. Όχι μόνο γιατί δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά, αλλά και για ό,τι έχουμε κάνει δεν φαίνεται να έχει γίνει αρκετά καλά. Ε, υπάρχουν ε, τράπεζες που με το ζόρι παραμένουν ζωντανές. Θέλω να αναφερθώ σε μία πτυχή ε, τη σχέση των τραπεζών με τις χώρες που τις διασώζουν. Υπάρχει ο εποπτικός μηχανισμός που προσπαθεί να λύσει βέβαια αυτό το πρόβλημα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Με την Order B και την εποπτεία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδήγησε η τράπεζα αυτή να διασωθεί με ελάχιστο κεφάλαιο χωρίς να ε, πτωχεύσει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου λοιπόν επέτρεψε να πάνε χρήματα σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις διάσωσης τραπεζών. Οπότε η ερώτησή μου είναι, πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός λειτουργεί, πιστεύετε ότι αυτή η διάσωση πάει πολύ μακριά γιατί διατηρούμε τελικά τράπεζες ζωντανές ενώ θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει σε καθάριση και πιστεύετε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου από τη δικιά του την πλευρά κάνει καλά τη δουλειά του, χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για το ποια τράπεζα είναι δημοσίου συμφέροντος και ποια όχι σωστά. Και μήπως τελικά αυτές οι τράπεζες απορροφούν υπερβολικά μεγάλα ποσά από το δημόσιο. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξει λοιπόν αυτό το πλαίσιο και να το προσπαθήσουμε εμείς από εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι το πλαίσιο εξυγίανσης θα μπορούσε να βελτιωθεί και θα μπορούσε να έχουμε πιο ισότιμους όρους. Τώρα από την άλλη μεριά η αφαιρεγκιότητα και η εναρμόνισή της, των κανόνων της δηλαδή, είναι κάτι το οποίο εξακολουθούμε να έχουμε στο τραπέζι. Πολύ θα ήθελα κι εγώ να δω πρόοδο για πολλούς και διάφορους λόγους. Όσον αφορά την εξασφάλιση καταθέσεων, γιατί υποθέτω ότι και αυτό θέλετε να ακούσετε, η πρόταση για διαφοροποίηση των σχετικών προγραμμάτων στη μεταβατική περίοδο χρειάζεται παρετέρω ανάλυση και σας ευχαριστώ που και εσείς συνεισφέρετε για τον στόχο μας να έχουμε μια πραγματική τραπεζική ένωση θα πρέπει να υπολογίζονται οι κίνδυνοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς για να ε, μειώνονται οι πιθανότητες κινδύνου. Η κάλυψη θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά να καταλήξουμε σε ένα πραγματικό έντις, εξασφάλιση καταθέσεων δηλαδή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απώλειες. Νομίζω ότι αυτές είναι οι ανησυχίες σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Μέλνταν από το ID. Ναι, καλημέρα. Θα μιλήσω γερμανικά. Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση στην ε, Γερμανία έχει ξεκαθαρίσει. Πλέον περιμένουμε η ΕΚΤ να συνεχίσει να επιτίθεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών μέσω χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων υποθέτω ότι ε, οι αντικοινωνικές αυτές ε, πολιτικές ε, θα συνεχιστούν. Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η πολιτική αυτή ουσιαστικά έχει αρνητικά, δημιουργεί αρνητικά κίνητρα. Και οι Γερμανοί και οι άλλοι βλέπουν τις καταθέσεις τους να εξατμίζονται. Λοιπόν, ε, θα πρέπει καλύτερα αντί να επικεντρωθείτε αποκλειστικά στην ορισματική ε, σταθερότητα να δείτε την πολιτική του κυρίου ε, Ντράγκη στο θέμα αυτό. Μιλήσατε για εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αυτή τη στιγμή τίνει προς το μηδέν. Δεν σας εμπιστεύεται κανείς και θα πρέπει να το γνωρίζετε. Έχετε κάποιες μελέτες ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να υπολογίζετε τον κίνδυνο της αρνητικής ε, κοινή ε, γνώμης για την ανήθικη πολιτική που ακολουθείτε. Έχετε κάποια ιδέα ή έχετε ερευνήσει σε ποιο βαθμό προχωράει η απαλωτρίωση των οικονομιών των ανθρώπων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους όπως τα κίτρινα γυλαίκα. Δεύτερη ερώτηση, πώς ε, μπορείτε να αναλαμβάνετε την ευθύνη για κάτι τέτοιο και σύντομο μικρόφωνο Και να έχετε ληστέψει 120 δισεκατομμύρια από τις οικοτομίες τους ε, και τρίτον, τι σκοπεύετε να κάνετε νομισματικά όσον αφορά το Green Deal ε, και τις υπόλοιπες ε, πολιτικές κομισιόν που θα συνεχίσουν να υπονομεύουν την οικονομία και τελικά να δημιουργήσουν ύφεση. Ε, με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Είπα ε, μέχρι δύο λεπτά οι ερωτήσεις. Αν έχετε την καλοσύνη, αφήστε την κυρία Λακάρτη να απαντήσει. Μία τελευταία πρόταση το δικό σας το whatever it takes τι θα είναι συγκεκριμένα, ποια μέσα θα χρησιμοποιήσετε εάν έχουμε ύφεση. Με συγχωρείτε, Κύριε Λαγκάρντα, έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε. καλημέρα σας. Ξέρετε, Νομίζω ότι όταν έχουμε περισσότερες δουλειές, ε, βελτιωμένη ανάπτυξη, ο πληθωρισμός είναι σε ένα επίπεδο που εγγυάται την σταθερότητα των τιμών, ε, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό είναι σύμφωνα με την εντολή που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όταν ε, το 2014 έλεγχαν μεγάλες αποφάσεις για να διευρυνθούν τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό έγινε για να στηριχθεί η οικονομία και να ανταποκριθεί η τράπεζα στην εντολή της. Οπότε δεν μπορεί να εστιάζεται σε μία πλευρά μόνο. Σε μια παρενέργεια την οποία αναφέρατε. Πρέπει να δείτε την γενική εικόνα και όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται και στο νομισματικό και στο δημοσιονομικό μέτωπο και από την σκοπιά των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και έτσι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει αυτά που έπρεπε. Τώρα, σαφώς. Θα ήταν ιδεώδες ε, και ε, οπωσδήποτε και εγώ θα ήθελα να περάσουμε σε ε, θετικά επιτόκια και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γιατί έχει ανέβει η παραγωγικότητα και η νομισματική πολιτική λειτουργεί ε, μαζί με την δημοσιονομική πολιτική. Αλλά πρέπει να κινηθούμε υπομονετικά για να κινήσουμε την οικονομία προς αυτήν την κατεύθυνση. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτά θα τα εξετάζουμε εκ του σύνεγγυς όταν καθορίζουμε την νομισματική μας πολιτική. Αλλά η νομισματική πολιτική πρέπει να αλλάζει σύμφωνα με τα γεγονότα που βλέπουμε, σύμφωνα με την εντολή που έχουμε και χωρίς ε, να τα κάνουμε χάλια για να είμαι Σας ευχαριστώ ο κύριος Γεκελούνας από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Λαγκάρντ όταν βγήκα βουλευτής ε, πριν από λίγους μήνες αναρωτιόμουν γιατί η επικοινωνία και οι μελλοντικέ κατευθύνσει είναι τόσο σημαντικές ε, για την Κεντρική Τράπεζα. Και βεβαίως αυτά τα ζητήματα συζητάμε σήμερα και την ε, οικονομική σταθερότητα. Και βεβαίως κοίταξα τον Οκτώβριο τα σχέδια της ΕΚΤ και είδα ότι σκοπεύετε ακριβώς να επεκτείνετε την έρευνά σας και στην οικονομική συμπεριφορά. Υπάρχουν και οι Άκελοφ Κάνεμαν και οι λοιποί νομπελίστες που έχουν ερευνήσει αυτά τα ζητήματα. Οπότε ίσως να αποτελούν αυτά ένα μέρος της απάντησης για να αντιληφθείτε και να διαχειριστείτε το οικονομικό σύστημα. Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο εργασίας ε, της ΕΚΤ του Καλ ε, που αφορά την ε, ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς ε, και βεβαίως οι βασικές λέξεις είναι ε, η ισορροπία η οποία επιτυγχάνεται, ο λεγόμενος ηθικός κίνδυνος, τα ζωικά ένστικτα κτλ. Ποιος είναι ο δικός ο ρόλος στην κατανόηση και διαχείριση αυτών των φαινομένων, γιατί για εμένα είστε κάποιο είδους ε, μάγο με κάποιον τρόπο πρέπει να διαχειριστείτε αυτά τα ζωικά ένστικτα μεταξύ άλλων να τα αναζωπυρώσετε όταν πρέπει ή να τα ηρεμήσετε ε, ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για αυτόν τον κλάδο των οικονομικών την έρευνα τη συμπεριφορά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ συγκεκριμένη και επίκαιρη ερώτησή σας. Εμείς ε, κοιτάμε περισσότερο τα νομισματικά και τα όσα γράφουν και οι μακροοικονομολόγοι. Αλλά σε μια προηγούμενη μου ζωή οπωσδήποτε ε, με απασχόλησε και το θέμα της έρευνας οικονομικής συμπεριφοράς ε, που σχετίζεται με την αποστολή μας. Οι συγγραφείς αυτοί βεβαίως βρίσκονται και αυτοί στην βιβλιοθήκη της ΕΚΤ και θα τους μελετήσουμε όπως και όλους τους άλλους. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχώς θέλω να καλωσορίσω τις ε, παουπηρές σας για βελτίωση της επικοινωνίας. Ο προκάτοχός σας ε, τα πέτυχε αυτό, απομονώθηκε ε, και μετά συγκρίθηκε μέχρι και με το κόμι Δράκουλα. Και το ίδιο και στη χώρα μου, η ΕΚΤ ε, ε, δεν χαίρει μεγάλης εμπιστοσύνης. Θεωρεί ο κόσμος ότι τον κλέβεται Εγώ ελπίζω ότι πραγματικά θα αυξήσετε τις, τις ικανότητές σας για να ακούτε τον κόσμο. Καλωσορίζουμε το πράσινο, το πράσινο σύμφωνο 11,5-3 ε, ε, ε, θα είναι το κόστος των επιπλέον κονδυλίων που θα χρειαστούν 3 εκατομμύρια τεράστια ποσά. Πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. να δούμε τι θα γίνει με την επανεξέταση της νομισματικής πολιτικής με ένα πράσινο QE. Ποιος θα το πληρώσει όλα αυτά τα ποσά. Ποιος θα πληρώσει την ύφη και ποιος είναι ο ρόλο της ΕΚΤ μέσα σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ναι, η πράσινη συμφωνία της Προέδρου, την οποία στηρίζει η Πρόεδρος Βαντελάγεν, είναι ένα project το οποίο προσωπικά καλωσορίζω και χειροκροτώ. Βέβαια όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους ε, και με την αποστολή που τους έχει ανατεθεί και σαφώς η ε, ΕΚΤ έχει μια ε, σαφή εντολή που έχει να κάνει με τη σταθερότητα των τιμών που εξαρτάται από ένα πλαίσιο που είναι πολύ καλά καθορισμένο και το οποίο θα αναθεωρήσουμε και μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής μας το 2020. Πώς μπορεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής να λειτουργήσει ως κομμάτι της, ε, της ε, επανεξέταση στρατηγικής μας. Αυτό θα το δούμε στους επόμενους μήνες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς σχηματίζονται οι σχετικές τιμές, οι, προ... Ε, εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, το πραγματικό κόστος, οι καταναλωτές αλλάζουν ε, συμπεριφορά και όλα αυτά είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις μετρήσεις μας και να ε, μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε και τις τιμές. Γι' αυτό λοιπόν, με βάση την αποστολή που έχουμε, αυτή, αυτές οι ε, Επιταγέ θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Τώρα, χωρίς βιασύνη, γιατί όπως είπα, πρέπει να έχουμε τα μέσα, τις μετρήσεις, να είμαστε σε θέση να δείξουμε πώς λειτουργούμε και ποια είναι ακριβώς τα μέτρα τα οποία ε, λαμβάνουμε. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε ποια είναι τα, τα collaterals για τις πολιτικές μας αυτές. Ε, οι κίνδυνοι να αξιολογηθούν σωστά. Η εποπτική επίσης λειτουργία της ΣΕΚΤ πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Μέσα σε αυτό το πνεύμα και αυτό το πρίσμα της εντολής της ΣΕΚΤ σίγουρα μπορούμε να συμβάλλουμε για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου που έχει εντοπίσει η σημερινή Επιτροπή υπό την ηγεσία της κ. Βαντερλάγεν ως επιτακτική ε, ανάγκη και ως επιταγή. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία, κυρία καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο, κάνατε μια αναφορά στην ε, ε, εξάπλωση του κορονοϊού. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, επειδή δεν αναφέρατε τίποτε ποσοτικό ως πρόβλεψη, ποια είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η επίπτωση στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομίας ή και της παγκόσμιας οικονομίας από την εξάπλωση του κορονοϊού. Έχετε κάποια σενάρια και κάποιες εκτιμήσεις γι' αυτό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας τις πείτε. Ε, η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τη χώρα μου την Ελλάδα. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε και από την προηγούμενη θέση σας, ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ελλάδα έχει βγει τον Αύγουστο του 2018 από τα μνημόνια έχει επιτύχει και το 19 και οι προβλέψεις και για το 20 είναι ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έχει εξασφαλιστεί μια σημαντική ελάφρυση του χρέους και έχει επανέλθει δυναμικά και με επιτυχία εδώ και κάμποσο καιρό και στην αγορά των ομολόγων. Η ερώτησή μου αφορά μια απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας που την περιμένουμε εδώ και καιρό. Το 2015 είχε μπει ένα όριο στην δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα. Οκτώ δις. Από τότε μέχρι τώρα η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά και το συνομολογείτε κι εσείς. Επομένως, να περιμένουμε σε αυτό μια θετική είδηση και μια θετική εξέλιξη. Και η δεύτερη μου ερώτηση. Πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή, η Επιτροπή μας ζήτησε με το σχετικό ψήφισμά της που θα συζητήσουμε και στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα να ενταχθούν και τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Πότε μπορούμε να περιμένουμε σε αυτό έναν οδικό χάρτη από την πλευρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρεστε σε περισσότερη ποσοτική χαλάρωση. Αποφασίστηκε το Σεπτέμβριο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο από ό,τι αποφασίστηκε το Σεπτέμβριο. Και είμαστε τώρα στο στάδιο υλοποίησης των όσων αποφασίστηκαν τότε που ήταν 20 δισεκατομμύρια μηνιαίως για το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο Πρέπει να δούμε την ε, καμπύλη μακροπρόθεσμα και κατά πόσο υποσχέσεις διατηρούνται. Νομίζω ότι όντως έχει επιπτώσεις και υπάρχουν και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και που αποφασίσαμε το Σεπτέμβριο. Τώρα να επικεντρωθούμε περισσότερο στο δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας που νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρη που έχει να κάνει με τα ελληνικά ομόλογα και το θέμα της επιλεξιμότητάς τους δεν είναι επιλέξιμα τώρα, σε αυτό το στάδιο του προγράμματός μας που ξεκίνησε 1η Νοεμβρίου της αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Και δεν είναι σε αυτό το στάδιο ούτε το 2015-2018 αν η κατάσταση συνεχίσει να βελτιώνεται, όπως συμβαίνει τώρα, και νομίζω ότι το είπε και ο συνάδελφός μου, ο αντιπρόεδρος Λουίς Ντεγκίντος, πριν από λίγες μέρες που ήταν για μια διάσκεψη στην Αθήνα, αν η κατάσταση συνεχίσει να βελτιώνεται και βάσει των κριτηρίων που εφαρμόζουμε σε όλες αυτές τις αγορές, πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι επιλέξιμα και τα ελληνικά ομόλογα. Γιατί υπάρχει σταδιακά βελτίωση. Και εδώ εκφράζω την ευχή να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί έτσι δείχνει ότι οι αγορές αξιολογούν την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ως συνεχώς βελτιούμενη. Οπότε βελτιώνονται και οι αξιολογήσεις. Ευχαριστούμε. Λίδια Περέιρα τώρα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Κύριε Λαγκάρντε, καλώς ορίσατε ε, και πάλι στο Κοινοβούλιο. Η δέσμευσή σας ε, ε, δείχνει και η προσήλωσή σας στις επαφές και στο διάλογο με την Επιτροπή μας δείχνει προμηνεί μάλλον αίσιες εξελίξεις όσον αφορά τη σχέση με το Εξήβριο Κοινοβουλίου και Κεντρική Τράπεζας. Ελπίζω και άλλοι θεσμοί να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα. Τώρα, για τις μη συμβατικές ε, πολιτικές ε, και κυρίως για τη διαδικασία ε, επανεξέτασης της στρατηγικής για την νομισματική πολιτική είναι καλά νέα και άμα ξεκινήσουμε με μια τόσο βαθιά συζήτηση όπως αυτή σημαίνει ότι συνεχίζουμε και εξετάζουμε όλες τις κατευθύνσεις λειτουργίας και άσκησης πολιτικής της νομισματικής πολιτικής. Η ερώτησή μου αφορά την εποπτεία. Η εποπτεία, η δημοσιονομική, μάλλον η οικονομική κρίση μας έκανε να πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερη εποπτεία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ανέβασε τους τόνους όσον αφορά αυτό όμως και συνεχίζουν να προκύπτουν σκάνδαλα ε, κεντρικές τράπεζες ε, όμως εξακολουθούν να επιλέγουν τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με το σημερινό σύστημα ε, τραπεζικής υποπτίας ή μήπως η κεντρική τράπεζα θα έπρεπε να είναι πιο δυσδυτική σε αυτό το τομέα. Πώς θα πείσετε τα εθνικά μέσα εποπτείας να χρησιμοποιούν κάθε δυνατότητα που έχουν γιατί δεν είναι μόνο μία ιδέα και μία αξία, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προστατέψουμε ε, για να αποφύγουμε τα σκάνδαλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Εποπτεία προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια διαφορά η οποία καθορίζεται από τα κατάοφλια τα οποία ε, φτάνουν ή όχι οι τράπεζες ε, ε, οι οποίες καλύπτονται από ευρωπαϊκή εποπτεία και αυτές που καλύπτονται από την εθνική εποπτεία. Και θυμάμαι συζητήσεις ε, με την ε, προηγούμενη επικεφαλής του Συμβουλίου Εποπτείας ότι πολλές φορές δίνονταν διαφορετικές ερμηνείες στην ίδια διάταξη. Υπάρχουν όντως εργαλεία και ολόκληρη η εργαλειοθήκη θα πρέπει να χρησιμοποιείται όσο γίνεται περισσότερο ώστε να παρεμποδίζονται αυτές οι πολλαπλές διαφορετικές ερμηνείες και τα κατόφλια που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες τράπεζες που ανήκουν στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης. Πιστεύω όμως ότι και στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης του ιστορμοκρατίας θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση. Καλύτερα ένας κανονισμός παρά οδηγία θα βοηθούσε πολύ σε αυτό το τομέα γιατί η, ε, εποπτεία ε, μπορεί να κυμαίνεται την πραγματική εποπτεία και συμμόρφωση προς ε, τις μακροπροληπτικές απαιτήσει και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, αλλά ε, μπαίνει και στα χωράφια των ε, και των εμβασμάτων που η, η Ευρώπη μπορεί να αυξήσει την εποπτεία που έχει ε, για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ η Έμιλι Ρέγνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του καιρού μας και κάθε δημόσιος φορέας πρέπει να συνεισφέρει για να γίνει η οικονομία τις επόμενες δεκαετίες κλιματικά ουδέτερη. Η ΕΚΤ ε, υποχρεούται από το άρθρο 107 της συνθήκης να στηρίζει τους ε, σκοπούς ε, της Ένωσης χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα των τιμών. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνεισφέρει στο στόχο αυτό η ΕΚΤ. Οπότε, η Κομισιόν υπολόγισε ότι θα χρειαστούμε 260 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο την επόμενη δεκαετία για να αποτελεμήσουμε αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή. Είναι διατεθειμένη η ΕΚΤ ε, να, να βοηθήσει να κινητοποιηθούν αυτά τα Και ο καθηγητής Βέλα είχε πει στο Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να σκεφτεί να δανείσει μεγάλα κονδυλία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα ίδια πιθανώς και αρνητικά επιτόκια τα οποία, με τα οποία δανείζει τώρα τις ε, τράπεζες ε, με αντάλλαγμα ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ε, και επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια στην Ευρωζώνη. Ε, θα κάνει κάτι τέτοιο η ΕΚΤ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, μια πολύ καλή ερώτηση γιατί με βοηθά να ξεκαθαρίσουμε το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μια υπηρεσία της Ένωσης οπότε δεν μπορούμε να δανείσουμε απευθείας σε αυτού χωρίς να παραβιάσουμε τη συνθήκη. Πρώτον, για παρόμοιου λόγου, ε, δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ομόλογα της ε, τράπεζα Επενδύσεων στην ε, πρωτογενή αγορά. Είτε μέσω δανείων είτε λοιπόν μέσω αγορά ομολόγων δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με τη συνθήκη. Η αγορά στην δευτερογενή αγορά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και έχουμε κάνει και στον βαθμό που η ΕΤΕΠ αυξάνεται σε όγκο, σε έκδοση ε, χρεογράφων κτλ. Οπωσδήποτε θα δούμε τις αγορές στη δευτεροκοινή αγορά των ομολόγων αυτών. Εκεί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι που νομίζω ότι είχα μόλις ανέφερα. Αλλά ε, δράτω τις ευκαιρίες να το ξαναπώ. αναφέρατε το πώς ε, η ΕΚΤ πρέπει να στηρίζει τους οικονομικούς στόχους. Περιλαμβάνουν διάφορα πράγματα και την ε, βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Ε, αυτό στηρίζουμε, δεν χαράζουμε εμείς την πολιτική. Είναι όλα αυτά υπό την αίρεση του βασικού στόχου, της σταθερότητας των τιμών. Αυτό το οποίο είπα και θεωρώ είναι ότι εντός του βασικού στόχου, η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος έχει έναν αντίκτυπο και πρέπει να συνυπολογιστεί. Επειδή έχει αντίκτυπο στις τιμές και τις σχετικές τιμές, στην κατανάλωση στους κινδύνους που αναμένουν οι καταναλωτές και οι εταιρείε. Και σχηματί είναι, συναποτελεί ένα από τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν ακριβώς υπολογίζουμε την σταθερότητα των τιμών που είναι η βασική μας εντολή. Είναι λοιπόν ένα διαφορετικό πρίσμα μέσω του οποίου μπορεί να και πρέπει να διοχετευτεί η βιωσιμότητα ε, του περιβάλλοντος για να καθορίσουμε σωστά τις τιμές και τον πληθωρισμό. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Γκαρθία Μαργάγιο. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα περιοριστώ σε γενικά ζητήματα, τα οποία όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Στα έγγραφα που έχουμε φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για ανησυχία. Υπάρχουν και πολιτικοί κίνδυνοι, όντως, όπως το είπατε κι εσείς, ε, στην αρχή κατάσταση ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα ήταν πολύ με μεγάλη ένταση και παραμένουν πολλά ε, ερωτηματικά ακόμα και για τη στάση των ΗΠΑ. Δεύτερον, για το Brexit, ούτε και εκεί είναι πολύ καλά τα νέα. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο νέος Πρωθυπουργό δεν θέλει τίποτα άλλο από ένα μοντέλο απλώς ελεύθερων συναλλαγών τύπου Καναδά. Δεν θέλει πιο στενές σχέσεις με την Ευρώπη. Και η κατάσταση για τις σχέσεις με το Ιράν επίσης είναι πολύ ανησυχητική. Ε, το θέμα της ε, στέγασης των ακινήτων. Επίσης είναι προβληματικό και οι το γνωρίζουμε πολύ καλά. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα σενάριο επιτάχυνσης όπως στην Ιαπωνία. Δηλαδή βρισκόμαστε χαμηλά στον πληθωρισμό, στα επιτόκια, με ανεργία όμως υψηλή σε μερικές χώρες, όπως για παράδειγμα στη δικιά μου. Κάποιοι εμπειρογνώμονες λένε ότι χρειάζονται δημοσιονομικά μέτρα είναι όμως πολύ περιορισμένα εξαιτία του μέγεθους του δημοσίου χρέους και επειδή οι νέοι κίνδυνοι, η ψηφιοποίηση και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτούν δύο πράγματα. Επενδύσεις και αντιστάθμιση στους διάφορους παραγωγικούς κλάδους. Αν είναι έτσι λοιπόν, ποια θα είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε αυτά τα πλαίσια από επιτάχυνσης την οποία ήδη την διαπιστώνουμε και η οποία απειλεί να επιδεινωθεί στο μέλλον. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Έχετε δίκιο για το ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι πολύ. Και όταν κάποιοι από αυτούς εξαφανίζονται, εμφανίζονται νέοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία μας και συμφωνώ μαζί σας για τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με το εμπόριο και τον εμπορικό κίνδυνο ΗΠΑ και Κίνας. Ναι, με αναβλήθηκαν, αλλά έχουμε άλλα νέα τώρα από την Κίνα για τον κορονοϊό και εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα και πώς θα επιδράσει την κινέζικη οικονομία αλλά και γενικότερα την παγκόσμια οικονομία. Οπότε και πάλι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να παρακολουθούμε και να έχουμε υπομονή. Τέτοιες πανδημίες έχουν την τάση να εμφανίζονται, να επηρεάζουν την κατάσταση, αλλά όταν εξαφανιστούν ανακάμπτει η οικονομία. Αυτό έχει συμβεί με το SARS, για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί εδώ η κατάσταση και πώς συνδέεται ε, με την ε, ε, διάδοση και πώς αυτή θα εξελιχθεί. Τώρα σε αυτό που περιγράψατε, χαμηλός πληθωρισμός, χαμηλά επιτόκια, χαμηλή παραγωγικότητα επίσης. Εδώ, ναι, είναι μια ανησυχία. Και ο λόγος που έχουμε την νομισματική πολιτική που έχουμε είναι ακριβώς γιατί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Όμω δεν θα σύγκρινα τη σημερινή κατάσταση της ευρωζώνη με την Ιαπωνία, με τίποτα. Η Ιαπωνία είχε μια περίοδο αποπληθωρισμού που κράτησε δεκαετίε, Οι προσδοκίε για τον πληθωρισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ήταν χαμηλότερες και είναι χαμηλότερες από ό,τι στην Ευρωζώνη, που είναι κάτω από το 1,7%. Συνεπώς είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση όπου ο πραγματικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία, αν λάβουμε υπόψη μας τον αποπληθωρισμό, είναι πολύ πιο ψηλός από ό,τι εδώ στην Ευρωζώνη. Συνεπώς δεν θα ήμουν τόσο αρνητική για την μακροοικονομική κατάσταση. Έχουμε δει κάποιες ενδείξεις σταθεροποίησης οι ενδείξεις και στη μεταποίηση είναι θετικές και είναι θετικές τους τελευταίους πέντε μήνες. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που είναι θετικές και πρέπει να στηριχτούν και να δείξουμε υπομονή και να στηρίζουμε την οικονομία ε, διατηρώντας το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Ευχαριστούμε. Έγινε Ρόγκλου τώρα. Ναι. κύριε Λαγκάρτ, χαίρομαι που είστε στην Επιτροπή μας ε, και συζητάμε τόσο τακτικά. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε λίγο περισσότερο και χαίρομαι για το ότι έρχεται πιο πολύ στο επίκεντρο του πολίτη, θα έλεγα, η ΕΚΤ, ε, για να αντιληφθούν και οι πολίτες περισσότερο την νομισματική πολιτική και να την έχουν κατά νου ε, και στις πολιτικές τους αποφάσεις. Ε, στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αφαιρθώ στον ισολογισμό της ε, ΕΚΤ. Έχουμε αυτή τη στιγμή φτάσει στα 4,5 3 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε ξεκινήσει με 720 δισεκατομμύρια το 2015, 2016 στα 916 δισεκατομμύρια μέχρι το 2018 που σταμάτησε η ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα και μετά ξανά 2019 το Νοέμβριο ξεκίνησε να αγοράζει κρατικά ομόλογα 20 ε, δισεκατομμυρίων κάθε μήνα. Οπότε ο ισολογισμός σας αυξάνεται συνεχώς και έτσι γίνεται όλο και πιο σημαντική η ΕΚΤ, παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο και εσείς προσωπικά άλλωστε γιατί έχετε μεγάλη θητεία. Οπότε το ερώτημα είναι προς τα πού πηγαίνουμε, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι αγορές και έχει γίνει δύσκολη η αναχρηματοδότηση των τραπεζών στην αγορά, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος παίκτης που τα αγοράζει όλα. και διαμορφώνεται έτσι το επιτόκιο ώστε να κερδίζουν τα ε, τα κράτη. Με ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια κράτη ε, εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την ε, ευκαιρία. Συντομεύεται, λέει ο Πρόεδρος. Για να αναδιαρθρώσουν το χρέος τους, αλλά άλλα δεν το έκαναν. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για τις χώρες αυτές. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η εντολή μας, ε, θα το λέω συνέχεια, είναι η σταθερότητα των τιμών και η νομισματική μας ε, πολιτική ε, ακριβώς έχει αυτόν τον στόχο. Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, τα προγράμματα αγοράς ομολόγων και αναχρηματοδότηση λαμβάνουν υπόψη δύο πράγματα. Πόσο αποτελεσματικό είναι και δεύτερον, τι κίνδυνο έχει. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κομμάτι του κινδύνου. Με ένα πλαίσιο ελέγχου κινδύνου όπου παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τους κινδύνους και όσον αφορά τώρα άγορες ομολογών ε, αγοράζουμε μόνο στοιχεία τα οποία έχουν επαρκή ποιότητα ορίζοντας όρια στον κάθε εκδότη για να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Είναι μια ερώτηση που ρώτησε και ο Έλληνα συναδελφό σα πότε θα είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα. Επειδή διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο και πρέπει να διατηρήσουμε το χαρτοφυλάκιο αυτό ασφαλές και στιβαρό, είμαστε πολύ προσεκτικοί και το παρακολουθούμε τακτικά αυτό για την σκοπιά του κινδύνου. Για την αποτελεσματικότητα είπα και να επαναλάβω ότι ο στόχος της σταθερότητας των τιμών έχει στόχο να στηρίξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ε, περαιτέρω ανάπτυξη, να στηρίξει τις επενδύσεις. Και ένας λόγος για τον οποίο η χρηματοδότηση των επενδύσεων, είτε μιλάμε από εταιρείες που αγοράζουν ε, νέο εξοπλισμό, μηχανολογικό, είτε νοικοκυριά όταν αλλάζουν ή αγοράζουν σπίτι ε, το κόστος χρηματοδότησης είναι χαμηλό τα τελευταία πέντε χρόνια ακριβώς λόγω της νομισματικής πολιτικής και από αυτήν την έννοια έχει βοηθήσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γκούναρ Μπέκ. Sorry about my technical incompetence. Αχ, με συγχωρείτε που δεν καταφέρνω να ανάψω το μικρόφωνο. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Θα τα πω καλύτερα γερμανικά. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Τον Σεπτέμβριο πέρσι συμφωνούσαμε όλοι ότι η ΕΚΤ υπό τον ε, προκατοχό δεν τηρούσε το γράμμα των συνθήκων και μας διαβεβαιώσετε και εσείς ότι και στο μέλλον δεν θα διστάσετε να παραβείτε τις συνθήκες ε, για το γενικό καλό. Ε, επιμένετε όμως τον στόχο του πληθωρισμού περί το 2% παρά το ότι δεν υπάρχει κάποια νομική βάση για αυτό. Λοιπόν, αυτή η φαινομενική αντίφαση μπορεί να ερμηνευθεί ε, ως εξής. Ε, οι στόχοι που θέτει από μόνη της η ΕΚΤ, όπως παραδείγματος ο πληθωρισμός 2%, είναι πιο δεσμευτικοί από τα όσα ορίζουν οι συνθήκες. Εάν ναι, γιατί. Εάν όχι, υπάρχει κάτι δεσμευτικό στις συνθήκες για την νομισματική πολιτική που θεωρείται εξίσου ε, σημαντικό όσο η ερμηνεία του Ντράγκη για την ε, νομισματική σταθερότητα να είναι 2% πληθωρισμός. Και δεύτερη ερώτηση. Με βάση το ΑΕΠ ε, της νομισματική της ε, ζώνης, η τράπεζα της Αγγλίας ε, έκδοσε γύρω στο 15% χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως έχει εκδώσει χρήμα ένα 40% του ΑΕΠ σε νόμισμα. Με τάση ανωδική. Δώστε μου σας παρακαλώ ένα ιστορικό παράδειγμα όπου το τύπομα χρημάτων μακροπρόθεσμα οδηγεί σε ανάπτυξη και οικονομική επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, όλα τα μέσα που έχει χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ ε, είναι εντός των ορίων της εντολής της. Ε, και στο παρελθόν Αυτά τα έχει επιβεβαιώσει και το δικαστήριο σε σχέση και με τις ε, απευθείας ε, αγορές αλλά και το πρόγραμμα αγορών δημοσίου τομέα πιο πρόσφατα όπου επίσης το δικαστήριο επανέλαβε την αναλογικότητα αυτών των μέτρων σε σχέση με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής. Ε, τώρα, αγορές ε, κρατικών ε, ομολόγων επίσης είναι σύμβατες με την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης του άρθρου 123 της συνθήκης. Οπότε, αυτές είναι οι νομικές παράμετροι και αποφάσεις του δικαστηρίου εντός των οποίων έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα. νομίζω οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές και οι όροι τους εξετάζονται πάρα πολύ προσωπικά από όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεύτερον, αναφερθήκατε στον στόχο του 2% και αναφέρθηκε και πιο πριν αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η σταθερότητα των τιμών το 1998 ήταν τότε ε, είχε τότε καθοριστεί ε, σε ένα πλαίσιο κάτω του 2%. Αυτό ήταν ο αρχικός ορισμός του 2098 και μιλάμε για εποχές όπου είχαμε τεράστιο πληθωρισμό σε σχέση με το σήμερα. Αυτή ήταν η αιτία λοιπόν, το ιστορικό. Το 2003 το πλαίσιο αυτό αναθεωρήθηκε ε, με μια, στρατηγική, με μια αναθεώρηση της στρατηγικής και ξέρετε, ανάμεσα στο 0 και το 2% υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο. Οπότε για να κατευθύνουμε τις προσδοκίες ε, καθορίστηκε στο κοντά αλλά κάτω από το 2%. Ε, επειδή ε, είπατε το τι κάνουν άλλες κεντρικές τράπεζες, αυτό λοιπόν είναι διαφορετικό από το τι κάνουν οι άλλοι. Είτε μιλάμε για την Τράπεζα της Αγγλίας ή το Fed όπως σας είπα είμαστε πολύ πιο κοντά στο 2% και είμαστε κοντά στο επίπεδο του ΦΕΔ της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω για να σας εξηγήσω τις παράμετρους, το πλαίσιο εντός του οποίου κινούμαστε. Και αυτό το πλαίσιο θα ξαναδούμε στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής. Οπότε, ε, σαφώς λειτουργούμε εντό της συνθήκης, ε, της εντολής μας ε, και της νομολογίας που μας δεσμεύει. Κοιτάξτε, και εγώ νομικός είμαι και ακολουθώ τους κανόνες, αλλά πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε πλήρως πάντα σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ. Πέντρο Σίλβα Περίρα. Σας ευχαριστώ κύριε Λαγκάρντα. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ε, κίνηση μιας τόσο σημαντικής επανεξέτασης της στρατηγικής ε, σε συμμόρφωση προς την εντολή της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και με την νέα πράσινη συμφωνία. Αλλά θέλω να σας συγχαρώ και για τα όσα δεν αλλάξατε. Ε, που στηρίζεται δηλαδή με τη νομισματική πολιτική στην οικονομική ανάπτυξη. Όμω η ερώτησή μου αφορά τη φορολογική πολιτική. Στην αρχική σα εισήγηση είπατε ότι ε, σε αυτή την περίσταση ήπιας ε, ανάπτυξης και όθησης και σας παραθέτω εδώ εσάς όχι μόνο η νομισματική πολιτική αλλά και η φορολογική πολιτική έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Βεβαίω αυτό δεν είναι κάτι το νέο ως αίτημα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς πώς εκτιμάτε την ε, ανταπόκριση της φορολογικής πολιτικής στην Ευρωζώνη της ε, δημοσιονομικής με συγχωρείτε, πολιτικής ε, στην Ευρωζώνη και πώς θα δράσετε αν η δημοσιονομική πολιτική δεν ε, ακολουθήσει αυτά που πρέπει για να εξασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη. Και επίσης ε, πώς ε, θα λειτουργήσουν εκείνοι που έχουν περιθώριο λιγμό όσον αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση. Είναι μόνο το μήνυμά σας αυτό μόνο για τη Γερμανία και την Ολλανδία ή πιστεύετε πως και άλλες χώρες έχουν περιθώριο λιγμού ώστε να κάνουν περισσότερα στην ε, δημοσιονομική τους πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας αυτή. Προσπαθούσα να σκεφτώ μια, ένα παραλληλισμό με τον αθλητισμό για να σας περιγράψω πώς πιστεύουμε πως η δημοσιονομική πολιτική που είναι σωστά σταθμισμένη μπορεί να ε, ε, ενισχύσει την νομισματική πολιτική και σκεφτόμουν ε, μια σκηταλοδρομία και πώς δίνει κανείς τη σκητάλη. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει, γιατί αν λειτουργούμε με σωστό συγχρονισμό, οι δύο πολιτικές βοηθούν ε, ε, η μία την άλλη. Η πολιτική υπεύθυνη για την δημοσιονομική πολιτική λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος της χρηματοδότησης είναι τόσο χαμηλό. Αλλά ε, και έχουμε πει και έχουμε υποδείξει σαφώς ότι Εκεί όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος θα ήταν σωστό ή οι θύνοντες για την χάραξη των πολιτικών να χρησιμοποιήσουν αυτό το χώρο για να στηρίξουν την οικονομία της Ευρωζώνης. Και δεν θα πω τώρα ακριβώς ε, ποιες είναι οι εν λόγω χώρες στον Ευρωζώνη που έχουν δημοσιονομικό χώρο. Απλά Θέλω να παρατηρήσω ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες που έχουν όντως δημοσιονομικό χώρο έχουν τώρα ξεκινήσει και χρησιμοποιούν αυτό τον χώρο για να στηρίξουν την οικονομία, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να επενδύσουν σε πράγματα που χρειάζονται. Και αυτό σίγουρα είναι ευπρόσδεκτο από τη δική μας προοπτική της ΕΚΤ, γιατί το να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στις επενδύσεις σε αυτές τις μακροχρόνιες ε, επιταγές που είναι η παιδεία, η σωστή ευρυζωνικό ίντερνετ, ένα σωρό πράγματα που είναι εργαλεία για το νέο περιβάλλον που θα καταστήσουν την ευρωπαϊκή μας οικονομία ισχυρότερη και πιο αυτόνομη, σαφώς ε, αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Ευχαριστούμε. Νταμία Καρέμου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Λαγκάρτ. Στην ακρόασή σα για το διορισμό σα, σα είχα ρωτήσει ποια θα είναι η σχέση σα με του πολίτε και χαίρομαι που σήμερα το πρωί δεσμεύετε υπέρ αυτή τη σχέση. Θέλετε η κοινή γνώμη να συμμετέχει, να τη ρωτήσετε ποια είναι η γνώμη τη. Μα εξηγήσατε τη θεματική πριν από λίγο. Ήδη όμως νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τα εκατομμύρια των πολιτών που κατεβαίνουν στους δρόμους ζητώντα να σώσουμε τον πλανήτη και ένα υπεύθυνο ε, σε επιχείρηση στη Γαλλία που λέει ότι δεν είναι μόνο το κλίμα, είναι και η οικονομία. Πάντα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλεγε ότι είναι ουδέτερη όσον αφορά τις αγορές για την αγορά ε, ενεργητικού από τις επιχειρήσεις. Τώρα με την επανεξέταση που θα κάνετε, θα ξαναδείτε και αυτή την αρχή και την εφαρμογή της, η οποία στην πραγματικότητα οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που καθ' άλλο παρά ουδέτερο είναι όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αγοράζει και που οδηγούν στον κλιματικό κίνδυνο. Η ΕΚΤ λοιπόν μέσω της εποπτείας της μπορεί να συνεισφέρει σε μια βιώσιμη οικονομία και να προστατεύει το περιβάλλον. Θα πάει και προς αυτή την κατεύθυνση η ΕΚΤ. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ναι. Θα σας πω περισσότερα, γιατί ξέρω, δεν φτάνει αυτό το ναι. Το πρώτο είναι αυτό που έθιξα και νωρίτερα με την κυρία Ρέγνερ, δηλαδή ποιος είναι ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην σταθερότητα τιμών και πώς ε, μπορεί να ληφθεί υπόψη καλύτερα. Σήμερα, εντάξει, τα νούμερα μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά αν δούμε τις 77.000 μελέτες που έχουν γίνει και έχουν δημοσιευθεί, αναλογικά θα δείτε ότι μόνο 0,1% έχει να κάνει με τα οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με το κλίμα, την κλιματική αλλαγή. Οπότε από πλευράς έρευνας ήδη Πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουμε περισσότερο για τη σχέση αυτή. Κλιματική αλλαγή, πληθωρισμός, κλιματική αλλαγή τιμές, κλιματική αλλαγή παραγωγικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή τα οποία μας ενδιαφέρουν στα πλαίσια της εντολής μας. Αυτή λοιπόν είναι η διάσταση έρευνας και ο αντίκτυπος των εργασιών αυτών ε, στην προσπάθειά μας για σταθερότητα τιμών που είναι και εντολή μας. Έπειτα, Υπάρχουν και κάποιες ε, βάσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρίς να αφισβητήσουμε την ουδετερότητα που αναφέρθηκε πριν. Μπορούμε κάλλιστα να δράσουμε. Ε, συνταξιδοτικά ταμεία, ε, ήδη πόροι της ΕΚΤ και για αυτά τα δύο, για τις επενδύσεις των συνταξιδοτικών ταμείων, για παράδειγμα, ήδη έχουν αναλυφθεί δράσεις και έχουν, έχουν δοθεί οδηγίες στους διαχειριστές και εξετάζουμε πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους δείκτες από δείκτες ουδετερότητας όσον αφορά τον άνθρακα και για τα αποθεματικά επίσης κοιτάμε πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα για την ε, νομισματική πολιτική αυτή καθεαυτή. Για τα διάφορα χαρτοφυλάκια κάπου το 80% είναι κρατικά ομόλογα, οπότε εδώ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και ένα 20% το οποίο αντιστοιχεί σε αγορά εταιρικών, ε, εταιρικού ενεργητικού. Αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε, ναι. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, το γνωρίζω και σε άλλες τράπεζες, κεντρικές τράπεζες, στο Διοικητικό Συμβούλιο επίσης. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει να το εξετάσουμε. Και έπειτα υπάρχει και όλη η πτυχή της πίστοσης, γιατί η εξασφάλιση ότι εξασφάλιση ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το εξηγούσα και νωρίτερα ότι προσέχουμε πάρα πολύ τον κίνδυνο και τον μετράμε ακριβώς για να προστατεύουμε το χαρτοφυλάκιο απέναντι στους κινδύνους. Αλλά οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή δεν λαμβάνονται ακριβώς υπόψη. Οπότε εδώ θα χρειαστεί μάλλον χρόνος ορίμανση των κριτηρίων αξιολόγησης να δούμε ποιου δείκτε θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν διάφοροι που αναδύονται σιγά σιγά, να δούμε αν θα τους χρησιμοποιήσουμε και κυρίως για διάφορες και κεντρικέ τράπεζες που έχουν προχωρήσει, το συζητάμε και ε, θα δράσουμε για να λάβουμε υπόψη μας τους κινδύνους. Δεν είμαστε όμως τώρα σε μια πολιτική σταθερότητα τιμών, αλλά διαχείριση κινδύνου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Φράνσε Φιτζέραλ τώρα. Ευχαριστώ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, κυρία Λαγκάρτ, και θέλω να καλωσορίσω τις διαπραγματεύσεις που θα κάνετε ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά το θεκιστικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό για όσον αφορά το τι αισθάνονται οι συμπολίτε μας. Τώρα είμαστε στην κατάσταση Brexit και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις, εμπορικές διαπραγματεύσεις σε ένα σύντομο διάστημα. Πώς πιστεύετε, να σας ρωτήσω, θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες το Brexit, ειδικά σε μια περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Και έπειτα, στενή συνεργασία ευθυγράμμιση με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις ε, δημοσιονομικές υπηρεσίες μετά το Brexit θα υπάρξει. Και έπειτα, και ε, ε, το θέμα του ορίου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 23%. Η ΕΚΤ έχει στην κατοχή της ένα σημαντικό κομμάτι ομολόγων Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και Γερμανίας. Ε, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ως ΕΚΤ ότι οι χώρες αυτές δεν θα επηρεαστούν δυσανάλογα από το 23% όριο έκδοσης και ότι το έκτε θα αγοράζει αυτό που δικαιολογείται. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσετε το όριο 23% στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης ή υπάρχουν περιστάσεις που θεωρείτε ότι μπορεί να προκύψουν όπου μπορεί να εξετάσετε την άρση αυτού του ορίου ή την αλλαγή αυτού κάποιες αντίξωες συνθήκες είτε σε μεμονωμένες χώρες ή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς για την ε, κατάσταση μετά Brexit. Να σας αναφέρω ότι εμείς στην ΕΚΤΕ είμαστε έτοιμοι. Έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ε, και ε, με την Τράπεζα της Αγγλίας έχουμε κάνει τις δικές μας ρυθμίσεις ώστε ε, τα νομίσματα και το ευρώ και η λίρα στερλίνα θα είναι διαθέσιμα και δεν θα ε, οδηγηθούμε, μάλλον δεν θα συμβάλλουμε σε περιόδους ρήξης ή ε, πτυτικότητας. σε, όλες τις, σε όλες τις γωνίες της, της Ευρωζώνης έχουν προειδοποιηθεί δε οι τράπεζες να προετοιμαστούν και να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όσον αφορά την ε, διαχωρισμό των σχέσεων το Δεκέμβριο, γιατί αυτό θα επηρεάσει κυρίως το εμπόριο. Τα θέματα τα δημοσιονομικά και τα τραπεζικά είναι χωριστά από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε τυχεροί που η Βασιλεία 3 εναρμονίζει, ε, μάλλον είναι μια πλατφόρμα εναρμόνισης υπό την οποία ρυθμίζονται οι τράπεζες σύμφωνα με την οποία εποπτεύονται και ελπίζουμε ότι το Brexit δεν θα είναι ευκαιρία για αγώνα προς τα κάτω και ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον που δημιουργεί η σύμβαση της Βασιλείας 3 θα τηρηθεί κατά γράμμα. Και στο πνεύμα της, μεταξύ δηλαδή των συμβαλωμένων μερών. Τώρα, η στενή σχέση που έχει δημιουργηθεί στη διάρκεια των ετών θα είναι διαφορετική. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να προχωρήσει στο Brexit δεν θα είναι η ίδια σχέση και δεν θα είναι ε, ε όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Λόγω της ε, διαφορετικής πρόσβασης, λόγω των διαφορετικών πληροφοριών, ελπίζω πως θα μπορέσουμε να έχουμε μία ε, παγιωμένη, σταθερή και καλή σχέση ε, παρότι θα απομακρυνθούμε, γιατί είναι προ το συμφέρον τη Ευρωζώνη να διατηρηθεί αυτή η σχέση. Τώρα, για το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης και το όριο πρέπει να σεβαστούμε την αναλογικότητα, πρέπει να σεβαστούμε τα κλίδες και τα όρια όπως ισχύουν και όπως προκύπτουν από τις ε, αρχές που είχαν εγκριθεί. Δεν θέλω να κάνω να σκεφτώ περίσταση όπου θα πρέπει να ε, προβλέψουμε ή να εξετάσουμε αν πρέπει κανείς ή να επιτραπεί η υπέρβαση των όρων, αλλά και σερά-σερά Θα το δούμε, θα πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε περίσταση και να ε, Είμαστε αποτελεσματικοί με βάση την εντολή που έχουμε υπό οποιαδήποτε περίσταση. Ελπίζουμε πως η, πολιτική μας θα είναι αποτελεσματική, ότι η δημοσιονομική αρχή θα είναι αρκετά δεκτική, ώστε να αποφύγουμε τέτοιες ε, περιστάσεις και καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ζωάν Βανόμπερφελτ. Ο Ζωάν Βανόμπερφελτ. Ευχαριστώ κυρία Λαγκάρντ. Έχω μία δήλωση και μία ερώτηση ε, θέλω να σχολιάσω και τη δήλωση. Η δήλωσή μου βασίζεται σε δηλώσει δύο συναδέλφων σα, τον κύριο Πανέτα και Μέσ. Ο κύριο Πανέτα είπε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τη ακροασή του τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρμοδιότητε για τη δημοσιονομική σταθερότητα γιατί αυτή είναι προπόθεση για τη σταθερότητα των τιμών. Και ο κύριος Μέσ ε, προσφάτως σε μια ομιλία στο Λουξεμβούργο είπε το εξή. Η αύξηση των τιμών ε, των ακινήτων και των λοιπόν στοιχείων ενεργητικού είναι υπερβολική και είναι ως αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά μεγάλης περίοδου ε, χαλαρής ε, νομισματικής πολιτικής. Λοιπόν, υπάρχει μια σιδηρή λογική εδώ πέρα, μια σιδηρά λογική. Η πολιτική νομισματική ανεβάζει τις τιμές των διαφόρων στοιχείων ενεργητικού που θέτει κινδύνο την σταθερότητα των τιμών. Οπότε ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτροχιάζεται από τον βασικό τη στόχο τη σταθερότητα των τιμών. Αυτή είναι η δήλωση που θα ήθελα να σχολιάσετε και η ερώτησή μου σχετίζεται με τι παρατηρήσει σα για την ψηλότερη παραγωγικότητα που βεβαίω ισχύουν και δικαίω τις κάνετε. Αλλά δεν συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να κολλάνε κεφάλαιο και εργασία σε ένα επίπεδο ώστε να επιζούν ως όφυλαν διάφορες οντότητες χάρη εντός εισαγωγικών στην πολιτική της ΕΚΤ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί, παρακολουθούμε την ε, οικονομική σταθερότητα και το κάνουμε αυτό σε όλα τα στοιχεία και η κύρια έντολή μας είναι η σταθερότητα των τιμών όχι ε, δημοσιονομική σταθερότητα αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε βεβαίως και η σχέση μεταξύ των δύο είναι κάτι το οποίο εξετάζουν πανεπιστημιακοί και πολιτικοί αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάποια στοιχεία μη ευθυγράμμισης ε, των διαφόρων ε, κατηγοριών στοιχείων στην Ευρωζώνη ε, λόγω των μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και δεν βλέπουμε σημάδια φούσκας στεγαστικής στην Ευρωζώνη στο σύνολό τους. Τώρα, υπάρχουν σε κάποια αστικά κέντρα οι τιμές των σπιτιών οι οποίες αυξάνονται ε, και οπωσδήποτε θα μπορούσαν οι τοπικές αρχές να εξετάσουν κάποια τοπικά μέτρα όταν δηλαδή δεν υπάρχει πρόσφορα ε, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, συζήτηση είναι μεγάλη ε, υπάρχει ένα ζήτημα τιμής που πρέπει να δούμε και να δούμε το θέμα της προσφοράς οπωσδήποτε. υπήρξαν κάποιες προειδοποιήσεις, θα θυμάστε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας τον Σεπτέμβριο του 2019 για το σημείο αυτό ακριβώς. Οπότε γνωρίζουμε τους κινδύνους ε, και προειδοποιούμε στο επίπεδο του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας. Τώρα, απειλεί αυτό το κατά πόσο είναι προσιτέ τιμέ ε, των ακινήτων. Πιθανώ γι' αυτό πρέπει να το δουν οι αρχέ, να δουν το, την πλευρά τη ε, προσφορά αλλά για την ώρα και έχω εκφράσει πολλές φορές την άποψή μου επ' αυτού η νομισματική πολιτική που έχουμε έχει σαφώς στόχο να διατηρήσει την σταθερότητα των τιμών να φτάσει στο επίπεδο που θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει τον στόχο μας ε, να στηρίξουμε την ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις. Και έρχομαι στη δεύτερη ερώτησή σας που σχετίζεται με το πώς συνεισφέρει η τράπεζα στην χαμηλή παραγωγικότητα μέσω του κόστου χρηματοδότησης που κάνει εύκολη τη ζωή στις μη παραγωγικές εταιρείε, ε, τις λεγόμενες εταιρείε zombie ε, που διευκολύνονται από την ε, χρηματοδότηση χαμηλού κόστους. Δεν βλέπουμε στοιχεία για κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να καταστήσουμε διαθέσιμη τη χρηματοδότηση και να ενθαρρύνουμε τη χρηματοδότηση επενδύσεων από όλου. Ανθρώπου, νοικοκυριά, από όλε τι εταιρείε και δεν μπορούμε να διακρίνουμε ε, μεταξύ μια εταιρεία η οποία δεν πάει καλά και δεν πάει καλά, δεν είναι η δική μα δουλειά. Εμεί ε, πρέπει να ε, διαθέσουμε χρηματοδότηση. Θα αναφερθώ σε μία μελέτη από την Δανία προσφάτως, όπου είναι αρνητικά τα επιτόκια πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι στην Ευρωζώνη. Και έγινε μία εμπειρική μελέτη, ότι δηλαδή η χρηματοδότηση δεν συνεισέφερε στην δημιουργία τέτοιων εταιριών ζόμπι. Σας ευχαριστώ. Τώρα, ο κύριος Έρο Λουόμα. Κύριε Λαγκάρτ, και εγώ χαίρομαι για την ε, ανακοίνωσή σας όσον αφορά τις προσπάθειες της ΕΚΤΕ για την επικοινωνία. Βέβαια, μια τέτοια προσπάθεια δεν θα πρέπει να συνίσταται μόνο στην εξήγηση της νομισματικής πολιτικής και ένα από τα σημαντικά στοιχεία εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να ενημερώνει το κοινό και για τους κινδύνους που ελοχεύουν στην Ευρωζώνη και στις αγορές. Ο Ντανιέλ Νόιμ, που ήταν πριν πρόεδρος του Παπτικού Συμβουλίου, είχε πει ότι ένας από τους βασικούς κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα της ε, Ευρωζώνης είναι ακριβώς το κίνδυνος από την νομοποίηση εσόδων ε, παράνομες δραστημιότητες. Συμφωνώ με αυτό. Και είναι κάτι το οποίο όντω είναι εντελώ απαράδεκτο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ευρωζώνη. Συγχρόνως γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το σκάνδαλο με τα μη ξυπηρετούμενα δάνεια απέκτησε κάπως κακή φήμη. Η ΕΚΤΕ θα έπρεπε να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Λοιπόν, ρωτάω πρώτον, θα μπορούσε η ΕΚΤ να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει αυτό ακριβώς το θέμα. Και το δεύτερο, από τη μακρά εμπειρία που έχετε, από τα χρόνια που ήσασταν επικεφαλής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γνωρίζετε ότι το αμερικανικό σύστημα ήταν, θα ήταν αρκετά ήπιο στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Τι έχετε να πείτε εσείς από την εμπειρία σας με το Αμερικάνικο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας για τα μη ξεπερωτούμενα δάνεια και για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την νομιμοποίηση ε, χρημάτων από παράνομες δραστηριότητε. Υπάρχει κατακαιρματισμός στην εποπτεία και επίσης ε, στον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου νομοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητε. Και αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα την περίπτωση των διασυνοριακών κεφαλαίων. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της παίρνει το θέμα πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά δεν είναι η έκτη που είναι υπεύθυνη για το ότι δεν προβλέπεται επαρκή νομοθεσία ή γιατί δεν χρησιμοποιείται το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την καταπολέμηση ε, της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν θα φτάσει για να αντιμετωπιστεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε στο τραπεζικό τομέα. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα κυρίως για τι διασυνοριακές δραστηριότητες. Συνεπώ, χαιρόμαστε πολύ για τις συζητήσεις που συνεχίζονται και είμαστε έτοιμοι να τις στηρίξουμε. Να προτείνω δύο πράγματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου θα βοηθούσαν να βελτιωθεί η καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και θα είναι πιο αποτελεσματικά τα μέτρα μα. Πρώτον, νομική βάση για να βασίσουμε τη δράση μα. Δεν νομίζω ότι η οδηγία η ευρωπαϊκή είναι ό,τι καταλληλότερο. Ευρωπαϊκό κανονισμό θα χρειαζόταν, γιατί τότε η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία είναι κάτι διαφορετικό και φαντάζομαι και η κυρία Νόη σε αυτό ακριβώ αναφερόταν στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν τα μέτρα στι διάφορε χώρε. Δεν θα υπήρχε αν είχαμε κανονισμό. Έπειτα, Χρειάζεται περισσότερο συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες αρχές που ασχολούνται με την υλοποίηση των μέτρων καταπολέμησης της νομοποίησης χρημάτων παράνομη δραστηριότητα και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η ΕΚΤ δεν έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση, για την εφαρμογή. Σίγουρα λείπει αυτό. Ευχαριστούμε. Η Ντανούτα Χούμπνερ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και σας άκουσα, κυρία Λαγκάρτα, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Γιατί ξέρετε ότι για ε, δεκαετίες το έχουμε αφήσει αυτό το θέμα στις δυνάμεις της αγοράς. Και εμείς ε, μπήκαμε ε, σε δεύτερη μοίρα, το ευρώ δηλαδή, ως διεθνές νόμισμα τώρα πριν από δύο χρόνια ο Σαν Κλοντ Γιούγκερ έθεσε το θέμα της ενίσχυσης του ευρώ στο διεθνές πλαίσιο και το έβαλε στην πολιτική ατζέντα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δύο ανακοινώσεις που μιλούν ακριβώς για την ενίσχυση του ευρώ. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ακόμα ότι οι δυνάμεις της αγοράς είναι αυτές που πρέπει να ασχοληθούν με αυτό ή ότι μπορούν να υπάρχουν και υποστηρικτικές πολιτικές. Επίσης, θυμάμαι ότι εσείς δεν έχετε μόνο την νομισματική πολιτική, έχετε και τα συστήματα πληρωμών. Οπότε μήπως και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Για την τελευταία θέλω να ασχοληθώ περισσότερο γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, το ευρώ το ευρώ είναι ένα από τα βασικά διεθνή νομίσματα. Ε, το εμπόριο γίνεται σε αυτό και όπως είπατε βρίσκεται στη δεύτερη θέση αλλά μακριά από το δολάριο. Αυξάνεται η αναλογία του στο καλάθι που έχει να κάνει με τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα και στην αναλογία αποθεμάτων που διακρατούν οι τράπεζες. Υπάρχει μια σταθερότητα, αλλά όντω βρίσκεται σε δεύτερη σειρά μακριά από το δολάριο. Τώρα, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ευρώ σημαίνει ότι υπάρχουν ε, ωφέλη, αλλά υπάρχουν και ευθύνε. Σίγουρα πάντως συνεισφέρει στην αυτονομία και στην ενίσχυση της περιοχής του κόσμου που εκδίδεται. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε τρει τομείς όπου πρέπει να συνεχίσουμε την πρόοδο και όπου ο δικό σας ο ρόλος είναι πολύ βασικός. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όπου το ευρώ να είναι ένα από τα δύο νομίσματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διεθνώ, τότε πρέπει να κάνουμε το εξή. Πρώτον, να μην έχουμε διεθνές ευρώ παρά μόνο εφόσον υπάρχει ε, κεφαλακή αγορά με ρευστότητα Χτες μίλησα γι' αυτό και πραγματικά με νοιάζει πολύ. Ιστορικά, αν δείτε, ένας από τους παράγοντες που βοήθησαν το δολάριο να ε, παραμερίσει τη στερλίνα ήταν η ρευστότητα της κεφαλαιαγοράς ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ένωση Κεφαλαιογορών πρέπει να γίνει πραγματικότητα και γρήγορα κυρίως με αυτά που συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή σκηνή και με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν αυτό δεν αποτελεί παράγοντα ώστε όλοι να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για την κεφαλαϊκή αγορά, ε, δεν βλέπω τι άλλο μας χρειάζεται. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχετε δίκιο που αναφέρεστε στα συστήματα πληρωμών. Πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά συστήματα πληρωμών αυτό στιγμή στην Ευρωζώνη και πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το TIPS, το σύστημα εκείνο που επιτρέπει η πρόσβαση ε, των τραπεζών στην ρευστότητα κεντρικών τραπεζών υπάρχει, πρέπει να διευρυνθεί και πρέπει επίσης και να έχουμε και ένα λιανικό σύστημα πληρωμών που να λειτουργεί καλύτερα, που να είναι ρευστό και που να το έχουμε φτιάξει εμείς εδώ. Και τρίτον, που είναι στοιχείο κλειδί είναι η ικανότητα που έχουμε να καταπολεμούμε τους κινδύνους στο κυβερνοχώρο. Δεν είναι μόνο θέμα αρχιτεκτονικής του συστήματος πληρωμών. Αυτά τα τρία, η Ένωση Κεφαλαγορών, συστήματα πληρωμών και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, είναι τρία στοιχεία στα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί αν θέλουμε πραγματικά το ευρώ να είναι διεθνές νόμισμα ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή, να σας πω ότι αυτά τα δύο θέματα είναι πολύ προσφυλή στην Επιτροπή μας. Μάλιστα, έχουμε ζητήσει εκθέσεις για την Ένωση των Κεφαλαγορών και για το Euro, ε, που είναι βέβαια υπό την έκρηξη του COP ε, για ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά γιατί όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι και είμαι ευτυχής που είχαμε έτσι την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Ο Ζήλ Μποαγιώ, τελευταίος ομιλητής, μετά λυπούμε αλλά δεν θα έχουμε χρόνο για το Catch the Eye γιατί έχουμε και μερικές ψηφοφορίε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λυπάμαι, δεν ήταν τελευταία ερώτηση, αλλά ειδου... Ε, ε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ και σας ευχαριστώ που θα μας υποδεχτείτε και στη Φραγκφούρτη. Ε, και ε, χαίρομαι που καταστήσατε την επικοινωνία προτεραιότητα. Η ΕΚΤ δεν είναι βέβαια ε, ο μόνος ευρωπαϊκός θεσμός που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Ευχαριστώ που όμως το ξεκινήσατε. Είναι περίπλοκα τα θέματα και εγώ ίδιος ακόμα είμαι όλος αυτιά για να μπορέσω να καταλάβω όλες τις επιτυχίες. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για τους αρνητικούς, τα, τα, τα αρνητικά επιτόκια. Πολύ εδώ εγκρίνουμε αυτή την πολιτική που κατά τη γνώμη μας είναι προσαρμοσμένη στις περιστάσεις και σύμφωνη με την εντολή που σας έχει ανατεθεί. Ωστόσο το γεγονός ότι πληρώνεται κανείς για να δανειστεί χρήματα είναι κάτι που διανοητικά είναι δύσκολο κανείς να το αντιληφθεί ε, και ε, όταν μιλάμε για ένα απλό πολίτη χωρίς να μπω στην τεχνική. Έχω δύο ερωτήσεις λοιπόν που τίθενται ως βουλευτής αλλά και ως πολίτης και ως φορολογούμενος. Θέλω να μιλήσουμε για τις πιθανές συνέπειες αυτής της πολιτικής. Καταρχάς επιτρέπει αυξημένη πρόσβαση στην πίστοση για τους ιδιώτες. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Διερωτώ με πώς οι τράπεζες θα αντισταθούν σε μία αύξηση επιτοκίων αφού έχουν δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ε, ενυπόθηκα δάνεια για, με πολύ χαμηλά επιτόκιο. δεν διατρέχουμε έναν κίνδυνο συστημικό ε, για τον τραπεζικό τομέα έτσι και ανεβάσουμε τα επιτόκια. Στη συνέχεια, τα πολύ χαμηλά επιτόκια μπορεί όντως να καλέσουν τους αποταμιευτές που δεν το ξέρουν όμως πάντα ε, να επενδύσουν σε πιο επικίνδυνα σε επενδύσεις για να αυξήσουν τα ε, χρήματά τους. Η επίτηση για αποδοτικότητα όμως δεν έχει μειωθεί και εδώ θα ήθελα να ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε αν γίνουν μαζικές ε, μετακινήσεις προς πιο επικίνδυνα μέσα Είμαι ένας απλός ευρωβουλευτής που προσπαθεί να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει για να μπορώ και με τη σειρά μου να το εξηγήσω στους άλλους. Ε, μην νομίζετε ότι ε, με κακή πρόθεση σε έτω αυτές τις ερωτήσεις. Ε, κύριε Λαγκάρτ, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που βλέπετε ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί ε, στην νομισματική πολιτική ήταν θεμητές και απαραίτητες για να στηριχθούν οι τιμές και να φτάσουμε αυτό το στόχο σταθερότητας των τιμών όπως ορίζεται από την εντολή της τράπεζας. Για τον πρώτο κίνδυνο που εντοπίζεται, δηλαδή το κίνδυνο τα νοικοκυριά να προστρέξουν με υπερβολικό τρόπο και να δανειστούν σε, με τρόπο ώστε να ε, είναι επικίνδυνο αυτό σε φάση που ξαναυξηθούν τα επιτόκια. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος και είναι ένας κίνδυνος ε, απέναντι στον οποίο ε, δύο μέτρα μπορούν να ληφθούν. Το ένα είναι μέτρα μακρο και μικροπροληπτικά, δηλαδή ε, τα όρια υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια ποσοστά, κάποιες αναλογίες που χρησιμοποιούνται, δηλαδή ποσό του δανείου σε σχέση με την ικανότητα ε, απόσβεσης, κόστος αγοράς σε σχέση με το επιτόκιο του δανείου και διάφορες τέτοιες αναλογίες και νομίζω μάλιστα οι Εθνικές Τράπεζες και, το, και η Τράπεζα της Γαλλίας θύμισαν ότι αυτά πρέπει να ε, τεθούν σε εφαρμογή. Και μάλιστα όσον αφορά τη διάρκεια του δανείου, γιατί διαπιστώνουμε και μία παράταση της ορίμανσης των δανείων. Και αυτό είναι κίνδυνος για τις οικογένειες που ε, παίρνουν δάνεια με χαμηλά επιτόκια και, σε, και πολύ μακροπρόθεσμα. Τώρα, τα μακρο και μικρό προληπτικά μέτρα, όπως σας είπα είναι αυτά. Δεύτερον, πριν από λίγο μίλησα για την απαραίτητη υπομονή Ελπίζουμε πως η μακροοικονομική κατάσταση όχι μόνο θα σταθεροποιηθεί αλλά σταδιακά θα βελτιωθεί και ότι η νομισματική πολιτική που τέθησε εφαρμογή και θα στηριχθεί και από μια καλή δημοσιονομική πολιτική θα επιτρέψει την ανάκαμψη της δραστηριοποίηση, την ανάκαμψη του ποσοστού πληθωρισμού και θα μας επιτρέψει να επανέλθουμε σε μια νομισματική πολιτική πιο ε, συμβατική ε, σιγά σιγά βέβαια είναι προφανές ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέσει να, να, να σπεύσουμε βραδέως ε, για να αποφύγουμε ε, το κίνδυνο για τα νοικοκυριά και για, για την οικονομία μας. Η ε, προσοχή και η φρόνηση θα πρέπει να βασιλέψουν όταν θα αλλάξει η κατάσταση. Τώρα, το σύστημα των δύο στρωμάτων τώρα που κάνει η αρνητική, τα αρνητικά επιτόκια να μην επηρεάζουν τις τράπεζες όταν μένουν μέσα στα συγκεκριμένα όρια που έχουμε θέσει και όταν αυτές τηρούν τα νόμιμα αποθεματικά. Τώρα, ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν κάποιοι θεσμοί ε, θα πρέπει να ε, προληφθεί και να χαλιφθεί από αυτού του ίδιου του θεσμού. Δεν είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι επενδυτικέ πολιτικέ, τι πολιτικέ hedging, οι διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και στον ε, ίδιο τον ορισμό των ε, στρατηγικών ανάπτυξη αυτών των θεσμών, ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ώστε να μπορέσουν να προβλέψουν του ενδεχόμενου κινδύνου. Πάλι θυμίζω ε, να είμαστε φρόνιμοι, να προχωρούμε ε, σιγά σιγά και μέχρι ότου βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η ακρόαση. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Λαγκάρντε που ε, ήρθατε και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Ένα λεπτό διάλειμμα μόνο θα έχουμε.